Καλημέρα σας. Τζιν Ντόμπρε στα πολωνικά. Και πολύ καλημέρα στα γερμανικά, στα γαλλικά. Θα ξεκινήσουμε. Θα συνεχίσω στα πολωνικά τώρα. Καλημέρα. Θα ήθελα να καλωσορίσω όλα τα μέλη της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μαζί με τους υπόλοιπους ε, προσκεκλημένους μας. Εγώ δεν έχω και πολλά να κάνω σήμερα το πρωί, αντιλαμβάνεστε. Απλά προεδρεύω της εκλογής ε, Προέδρου της ε, Υποεπιτροπής μας για το δεύτερο μισό της θητείας αυτής και κυρίες και κύριοι με ενημερώνουν πως η κυρία Λοχμπίλερ είναι η υποψήφια για ε, πρόεδρος και στο δεύτερο μισό της ε, θητείας. Υπάρχουν άλλες υποψηφιότητε. Ο κύριος Ταβάρες. Well, uh, I have nothing else to say Then... Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Ο κυρία Λόχ Μπίλερ θα είναι εξαιρετική πρόεδρος της Επιτροπής και χαίρομαι για αυτή την απόφαση. Ε, Μάλιστα, κύριε Δόμσκης. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ τα ίδια. Και οι φιλελεύθεροι θέλουν να εκφράσουν ε, την εκτίμησή τους στην Μπάρβαρα Λόχμπίλερ και θα την υποστηρίξουμε. Μάλιστα. Τα ίδια και οι φιλελεύθεροι. Κύριε Χάουιτ. Πρέπει όλοι να μιλήσουμε λοιπόν, θα τα πω κι εγώ. Αλλά ειλικρινά σας λέω πως ε, η Μπάρβαρα Λοχμπίλερ ήταν ε, εξαιρετική πρόεδρος και θα ήταν ε, σοκ εάν δεν ήθελε να συνεχίσει. Να παρακαλώ στους πράσινους, ε, μας έχετε δώσει μια εξαιρετική πρόεδρο, μην την αλλάξετε. Ευχαριστώ και η κυρία Βέιντερ. Ναι, και από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και εμείς τα ίδια θα λέγαμε. Και ανησύχησα και έλεγα πω πω Θεέ μου να μην φύγει η κυρία Λοχμπίλερ. Αλλά ευτυχώς θα συνεχίσει και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Ακούτε λοιπόν εν χορό τους συναδέλφους, τις πολιτικές ομάδες, οπότε μπορούμε να εκλέξουμε την κυρία Λοχπίλερ διαβοής. Συγχαρητήρια, κυρία Λοχμπίλερ. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω λοιπόν να έρθω να καταλάβετε τη θέση της Προέδρου και να σας πω πως είμαι σίγουρος πως η κυρία Λοχμπίλερ θα κάνει εξαίρετο έργο. Uh, Ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε. Μου αρέσει η δουλειά στην ε, Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και νομίζω πως ε, από τον Σεπτέμβριο που κάνω αυτή τη δουλειά. Ε, την απολαμβάνω γιατί ολόκληρη η Επιτροπή δουλεύει ως μια ομάδα και είμαι πεπισμένη πως ε, θα συνεχίσουμε έτσι με αυτό το συναδελφικό τρόπο λειτουργία. Τώρα περνάμε λοιπόν στην εκλογή του, των αντιπροέδρων. Περνάμε λοιπόν πρώτα στην εκλογή του πρώτου αντιπροέδρου. όλες οι πολιτικές ομάδες συμφώνησαν να προτείνουν τον κύριο Ζιμπ ο οποίος ε, ήταν αντιπρόεδρος ε, και στο παρελθόν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητε. κύριε Τούκες την ε, κυρία Ενιές Λεμπρούν θα ήθελα να προτείνω για δεύτερη αντιπρόεδρο. Ευχαριστώ. Και είστε υπέρ του κυρίου Ζιμπ. Ναι, ναι, βεβαίως. Βεβαίω, ναι, το ΕΛΚ στηρίζει τον κύριο Ζιμπ. Μάλιστα, κάποιο άλλο. Κύριε Ντόνσκι. Ναι, κύριε Πρόεδρε, Εμείς από το ΑΛΤΕ προτείνουμε τον κύριο Καζάκ ε, ως αντιπρόεδρο. Και για τρίτη, τρίτη αντιπρόεδρο, τέταρτη μάλλον, με ενημερώνουν πως είναι η κυρία Ιωάννα Σένισιν. Υπάρχουν ε, άλλοι υποψήφοι. Κύριε Χάουιτ. Ναι, είναι θετικό όταν έχουμε συναδέλφους ε, που έχουν καταλάβει ήδη τα αξιώματα να συνεχίζουν, αλλά καλό είναι το ότι επεκτείνεται και η Επιτροπή μας βεβαίως με νέους συναδέλφους όπως με την κυρία Σέτσιν η οποία θα παίξει ένα πολύτιμο ρόλο τώρα στην υποεπιτροπή μας και την είμαι ικανοποιημένος που μπορώ να την καλωσορίσω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, οπότε οι υποψηφιότητε που έχουμε είναι ο κ. Ζήμπ για πρώτο αντιπρόεδρο, η κυρία Λεμπρούν για δεύτερη αντιπρόεδρο. Δεν είναι εδώ νομίζω. Εντάξει. Ο κύριος Καζάκ για τρίτος αντιπρόεδρος και τέταρτη η κυρία Σεντσίν. Υπάρχουν άλλες υποψηφιότητε. Όχι. Νομίζω λοιπόν πως μπορούμε να τους εκλέξουμε διαβοής. and I would like uh, to ask you to... Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να καταλάβετε τις θέσεις σας εδώ στο Προεδρείο. Επίσης, να ευχαριστήσω όσους ε, διατέλεσαν την πρόεδρη και νομίζω κάποιοι θα συνεχίσουν κιόλας, κυρία Αντρικένη. Yes. Ah, okay. So, then uh, again it's a little bit late, but I wish. Μάλιστα, να ευχηθώ και καλή χρονιά μια που είναι η πρώτη μας συνεδρίαση φέτος και ελπίζω ε, η δουλειά μας να οδηγήσει σε πραγματική βελτίωση της δύσκολης κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, όπου και αν αυτή υπάρχει. Και Σήμερα βεβαίως έχουμε μια πλήρη συνεδρίαση και ως συνήθως ε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ρωτήσω αν εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Θέλετε να προσθεθεί κάτι. Όχι, άρα εγκρίνεται. Και βεβαίως έχουμε αποστείλει και το πρόγραμμα Έχουμε αποστείλει τα πρακτικά του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου. Εγκρίνονται. Ωραία, σας ευχαριστώ. Περνάμε λοιπόν στις ανακοινώσεις της Προέδρου. Μετά λοιπόν την απονομή του βραβείου Ζαχάροφ είχαμε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση και ομιλίες με τους ε, ε, βραβευθέντες και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην περιοχή όπως κάναμε και στο παρελθόν. Θα εστιάζουμε λοιπόν σε κάθε χώρα, σε μία χώρα σε κάθε συνεδρίαση και θα δούμε τι γίνεται στις αραβικές χώρες. Πριν τα Χριστούγεννα και ε, την Πρωτοχρονιά στην Αίγυπτο πάταξαν θα έλεγα τις ΜΚΟ εθνικές και διεθνείς και πρέπει να πούμε στις Αιγυπτιακές αρχές πως αυτό μας ενοχλεί ιδιαίτερα και πως θα πρέπει να σταματήσουν να προκαλούν τις ε, ΜΚΟ και νομίζω πως ε, αυτό έχει σχέση και με την νομοθεσία η οποία είναι περιοριστική για μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Τώρα, η Aung η οποία το 1990 είχε βραβευτεί με το βραβείο Ζαχάροφ. Φαντάζομαι θα μάθατε πως ε, ε, στη χώρα της υπήρχαν θετικές ε, εξελίξεις και ελπίζουμε αν βελτιωθεί η κατάσταση να μπορέσει να έρθει στις Βρυξέλλες και να παραλάβει αυτό προσώπο στο βραβείο της. Τώρα η κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία Βυρμανίας Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πάει στη χώρα αυτή τον Φεβρουάριο και αυτό νομίζω πως είναι καλό γιατί Υπάρχουν πολλές προκλήσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καλό θα ήταν ε, να, υπάρξει και κάποια συνοδεία από την από την Επιτροπή ε, Δικαίου ε, Νομικών Υποθέσεων και καλό θα ήταν να ταξιδεύουμε και εμείς μόνοι μας ε, για να συναντηθούμε και με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου της χώρας αυτής. Τα ζητήματα βέβαια αφορούν τις εκλογές, πολιτικούς κρατούμενους, κρατούμενους συντήρησης, παιδική εργασία και τα λοιπά. Επίσης είχαμε την 11η επέτειο της σύστασης ε, του Κέντρου Κράτησης του Γκαντανάμου. Συνολικά 779 κρατούμενοι ε, πέρασαν από εκεί, 171 παραμένουν και το έτοιμά μας είναι βεβαίως η κυβέρνηση των, η επανακλήση το κέντρο αυτοκράτησης και οι άνθρωποι οι οποίοι κρατούνται να δικαστούν και αν δεν γίνεται αυτό να αφαιθούν ελεύθεροι. Δυστυχώς δεν έχει υπάρξει κάποια αλλαγή, τα πράγματα έχουν χειροτερέψει γιατί με, την με το νέο στρατιωτικό δόγμα είναι ξεκάθαρο πως δεν θα μεταφερθούν στην επικράτεια των ΗΠΑ οι κρατούμενοι οπότε δεν θα μπορέσουν να δικαστούν σε μη στρατιωτικό δικαστήριο στην Κίνα. Τις τελευταίες εβδομάδες οι κινέζικες αρχές αύξησαν την πίεσή τους, καταδίκασαν πάρα πολλούς δικηγόρους και διανοούμενους σε ποινές ε, με την κατηγορία του ότι υποκινούν την ανατροπή του καθεστώτος Ο Τσεν καταδικάστηκε σε φυλάξη 9 ετών το Δεκέμβριο και ο Τσένξι σε φυλάξη 10 ετών με τις ίδιες κατηγορίες. Ο Ζου Γιουφού, ένας ποιητής, συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες, ενώ ο συγγραφέας και ακτιβιστής Λίτη επίσης καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλακή. Επίσης, ο Χουτζία, που είχε λάβει το βραβείο Ζαχάροφ το 2008, ανακρίθηκε από την αστυνομία ε, για πολλές ώρες στις 12 Ιανουαρίου. Είχε αποφυλακιστεί ούτως ή άλλως ε, πέρσι τον Ιούνιο, αλλά περιορίζονται οι δραστηριότητες του ούτως ή άλλως από την απόφαση του δικαστηρίου. Η αντιπροσωπεία μας λοιπόν που θα πάει στην Κίνα ε, της ε, Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων συνομίλησε με την αντιπροσωπεία για την Κίνα και είπαμε πως στην επόμενη συνεδρίασή τους θα πάω και εγώ να τους μιλήσω για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οπότε... Δεν ξέρουμε πώς θα γίνει αυτό. Είχαν ορίσει μια ημερομηνία το Δεκέμβριο. Απλά δεν ήμασταν σίγουροι. Τώρα για τη Ρωσία. Έχουμε θετικά νέα θα θυμάστε επίσης ε, την οργάνωση βραβημένη βραβείο Ζαχάροφ ε, την Memorial ε, ο επικεφαλής ο οποίας ο Όλε Γκορλόφ απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες που οποίες αντιμετώπιζε γιατί άλλαξε η νομοθεσία όσον αφορά τη δυσφήμιση γιατί είχε κατηγορηθεί γιατί κατηγόρησε δημόσια τον Τσετσένο πρόεδρο Καντήροφ ως πολιτικά υπεύθυνο για την δολοφονία της ε, Ναταλίας ε, Στεμίροβα, μέλους της οργάνωσής του, πριν από ένα έτος. Τα αρνητικά όμως είναι πως υπάρχει ακόμα μία υπόθεση στα δικαστήρια για ε, αποκάλυψη κρατικών μυστικών μια υπόθεση που ξεκίνησε μετά από μήνυση της πολιτοφυλακής της Τσετσενίας κατά του κυρίου Ιγκόρ Καλιάπιν, που είχε επίσης βραβευτεί το 2011 και είναι επικεφαλής της μικτής κινητής ε, ομάδας της Τσετσενίας που ερευνά παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οπότε εμείς προτρέπουμε τις ρωσικές αρχές να μην παρενοχλούν τον κύριο Καλιάπιν για στην δουλειά του, η οποία είναι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και νομίζω πως ε, θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στη Ρωσία και σας υπενθυμίζω πως στις 8 Φεβρουαρίου έχουμε και μία ακρόαση. Τώρα για τη Λευκορωσία. Κάποιοι από εσάς και από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ήρθαν σε μια συνάντηση που είχαμε χθε μαζί με την αντιπροσωπεία για τη Λευκορωσία και την υποεπιτροπή μας και εκεί πέρα μας μίλησαν τρεις ΜΚΟ για την κατάσταση στη Λευκορωσία. Ήταν σαφή το ότι η κατάσταση επιδεινώνεται και ιδιαίτερα θα πρέπει να αυξήσουμε την πίεση, την οικονομική στην κυβέρνηση Λουκασέγκο ίσως μέσω της πίεσης διαφόρων ε, εταιριών. Το εξετάζουμε αυτό. Το πώς μπορεί να γίνει. Επίσης, είχαμε και τη μητέρα του Βλάντισλαβ Καγιάλεφ, ε, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε θάνατο. Ήταν η μητέρα του εδώ πέρα. Και μας συζήτησε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο για την περίπτωσή του. Η κυρία Βαϊντέρη λοιπόν έκανε την πρόταση να απευθύνουμε μία επιστολή στον πρόεδρο Λούκασέγκο να δώσει χάρη στον άνθρωπο αυτό. Σας υπενθυμίζω πως ε, ε κατηγορεί το ότι συμμετείχε στην ε, επίθεση στο μετρό του Μίνσκ μία κτηνώδη επίθεση και βεβαίως ε, στη Λευκορωσία ε, όταν κάποιος έχει καταδικαστεί σε θάνατο δεν ε, ενημερώνονται οι οικοί του για το πότε θα γίνει εκτέλεση. Και ευτυχώς ο νέος μας πρόεδρος, ο κύριος Σούλτς, ε, έκανε μία δήλωση επευθυνόμενος προς τον Λουκασέγκο και αναφέρθηκε και στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση. Οπότε, όπως έγραψα και για το Δεκέμβριο, και είχα απευθύνει μια επιστολή ούτω ή άλλω. Ε, δεν νομίζω πως χρειάζεται να το επαναλάβουμε γιατί ήδη ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου το έκανε. Απλά ζήτησα από το προσωπικό τη Επιτροπής ε, να προετοιμάσουν μια επιστολή για δύο άλλες περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν επίσης καταδικαστεί σε θάνατο. Αυτό θα το δούμε με τις πολιτικές ομάδες. Θα το δούμε και με βάση τις εκλογές το Μάρτιο στη Ρωσία. Θα επιταχύνουμε και με το θέμα της Λευκορωσίας, διότι θα ζητήσει υποστήριξη η Λευκορωσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι από τους Ρώσους. Άρα θα είμαστε σε επαφή με την αντιπροσωπεία της Λευκορωσίας για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να εκδώσουμε ένα ψήφισμα. Ως προς τις σημειώσεις της Προέδρου, προσπαθώ να μην εστιάσω την προσοχή μου σε συγκεκριμένες περιφέρειες και δεν είδαμε την Λατινική Αμερική μέχρι τούδε. Βεβαίως θα έχουμε μια κρόαση με την Λατινική Αμερική σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά τη Δευτέρα ο πρόεδρος του Έλσαλβαντόρο, ο κύριος Φούνες, ζήτησε για πρώτη φορά συγνώμη στο λαό του για ε, μια γενοκτονία στην ουσία του στρατού 30 χρόνια πριν. Μεταξύ 11 και 13 Δεκεμβρίου του 1991 και ο πρόεδρος ε, είπε ότι αυτή η σφαγή είναι στο Ελμοσότε και είναι και η μεγαλύτερη σφαγή μέχρι τώρα. Επρόκειτο κατά τη, για τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, αλλά κατά τη διάρκεια αυτής της σφαγής σκοτώθηκαν πολλοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 460 παιδιά. Είναι εξαιρετική σημασία στο γεγονός ότι ο πρόεδρος ζήτησε συγγνώμη δημοσία και από το μάλλον μέχρι το 1992, ο Εθνικός Στρατός στο Ελσαλβαδόρ, καθώς και η κυβέρνηση αρνήθηκαν ότι η σφαγή είχε λάβει η χώρα μόνο όταν οι ατροδικαστές από την Αργεντινή ανέλαβαν έργο και κατά τη διάρκεια ανασκαφών βρήκαν αποδεικτικά στοιχεία για τη σφαγή. Και δυστυχώς οι υπεύθυνοι δεν έχουν διωχθεί. Άρα ευτυχώς καταπολεμάται η ατιμορρησία. Ως προς την Αφρική, είπα πολλές φορές ότι στην, ε, στα θέματα μας θα πρέπει να συζητηθεί και η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αφρική. Ο κύριος Τόκες επίσης ε, μας μίλησε για την κατάσταση στην Ιγυρία. Το είδαμε και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. δηλαδή το Boko Χάραμ που σημαίνει ότι η, δυτική, η εκπαίδευση δυτικού τύπου απαγορεύεται, ε, έχει διωχθεί και είναι κάτι το οποίο είδαμε και στα ΜΜΕ. Και επειδή οι διωκόμενοι είναι μουσουλμάνοι χριστιανοί και η αστυνομία, η δίωξη και η σύραξη μάλλον αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αναμενόταν. Εμπλέκονται και τα Ηνωμένα Έθνη. Γι' αυτό θα ήθελα εσείς και οι πολιτικές ομάδες να δείτε πόσο μπορείτε να συντάξετε ένα ευρύτερη εμβέλειας ψήφισμα για την κατάσταση στην Ιγυρία ως προς τα διάφορα θέματα στον, στην αναθεώρηση της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Λέδη Άστον μας μίλησε για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δημοκρατίας, που βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της ΕΙΕΔ. Έτσι αναθεωρούμε τα, την πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λάβαμε αυτό το έγγραφο. Μετά από μια διευρυμένη συζήτηση συμφωνήσαμε ότι η επόμενη έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα αφορά μια ανακοίνωση για την αναθεώρηση αυτή. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε στο διευρυμένο Προεδρείο, διότι όταν βλέπω τις συζητήσεις στα κράτη-μέλη για ότι και ε, ο Δανός Υπουργός Εξωτερικών μας μίλησε για τις απόψεις του. Άρα μέχρι το τέλος της Προεδρίας της Δανίας θα μπορούσαμε να έχουμε ένα διευρυμένο, μια διευρυμένη αναθεώρηση και σύνθετη καθώς και συνεκτική έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια συνένεση ή μια κοινή δήλωση από όλα τα θεσμικά όργανα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για να δούμε ποια είναι τα πιο βασικά ζητήματα για μας. Παράλληλα, η κυρία Μαρινάκη θα συζητήσει μαζί μας αυτό το θέμα. Ε, δυστυχώς όμως δεν μπορεί να βρίσκεται μαζί μας και άρα στις 9 Φεβρουαρίου με τον κύριο Ποπόφσκι θα το συζητήσουμε και ελπίζω να μπορέσουμε να εργαστούμε επί της ουσίας, γιατί στο διευρυμένο Προεδρείο θα πρέπει να ξέρουμε ποιος θα εργαστεί σε αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας και θα πρέπει να ληφθεί μια συνενετική απόφαση. Ως ε, τον κανονισμό για την αντιμετώπιση του βασανισμού θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι του, στο εμπόριο, στις εμπορικές συναλλαγές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό αφορά και τις ε, διάφορες ενέσεις ε, τα αναισθητικά που χρησιμοποιούνται, τα ναρκωτικά που χρησιμοποιούνται στις ενέσεις ε, για την επιβολή της θανατικής ε, ποινής στις χώρες που δεν έχουν καταργήσει τη θανατική ποινή. Χαιρόμαστε λοιπόν ότι, γιατί η Επιτροπή έδρασε αμέσως επί του θέματος αυτού και θα ήθελα να πω ότι λέει Άστον ότι όταν σχολίασε αυτή την απόφαση μίλησε για την αντίταξή μας στην θανατική ποινή και μίλησε για την απαγόρευση εξαγωγής αυτού του αναισθητικού. Είναι το πρώτο βήμα για να ανταποκριθούμε στις εκκλήσεις της κοινωνίας των πολιτών για να ενισχύσουμε την δική μας νομοθεσία. Και τον επόμενο χρόνο θα αναθεωρηθεί και η σχετική νομοθεσία. Όπως ξέρετε, είχαμε μία συζήτηση εδώ στην υποεπιτροπή μας, διότι υπήρχαν και άλλα τέτοια ε, προϊόντα τα οποία είχαν εξαχθεί, όπως ε, χρήση ηλεκτροσόκ και ειδικά... So, uh, uh, και ειδικέ χειροπέδες που ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνες στη ε, χρήση τους. Ο κύριος Χάουιτ θα ήθελα να πω ότι ενισχύουμε και δεχόμαστε αυτά που είπατε σε σχέση με το διευρυμένο Προεδρείο και αυτά που είχαν συζητηθεί έγινε ένα συμβιβασμός με βάση τα στρατηγικά στοιχεία αυτής της έκθεσης. Υπήρχε ένα προσχέδιο ε, προβλέπω μία μικρή παράγραφο για τις ε, κυρώσεις και θα υπάρξει και ένα ε, ψήφισμα με βάση αυτά που συμφωνήθηκαν στο διευρυμένο Προεδρείο και νομίζω ότι θα πρέπει να επισυναυθεί. Ευχαριστούμε Ρίτσαρτ Χάουερτ που μας το υπενθύμησες και όπως ξέρετε θα προβλέψουμε χρόνο για αυτή την έκθεση στην επόμενή μας συνεδρίαση. Υπάρχουν άλλα σχόλια παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επανέλθω στο ζήτημα, λέει η κυρία Βάιντερε, στο ζήτημα αυτό που θίξατε, γιατί όταν, ε, μάλλον, όταν συναντηθήκατε με αντιπροσωπεία της Λευκορωσίας, με την αντιπροσωπεία της Λευκορωσίας, ακούσατε πολλά. Ακούσαμε ε, αρκετά και για τη θανατική ποινή, Υπάρχει λοιπόν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία. Αυτοί οι νέοι άνθρωποι που έχουν καταδικαστεί με βάση πολύ ε, αδύναμα στοιχεία, αν μπορούμε να τα αποκαλέσουμε καν στοιχεία, με βάση αυτά τα ελλειπή στοιχεία, δεν θα έπρεπε να καταδικαστούν διότι γνωρίζουμε ότι οι περισσότεροι είναι αθώοι. Νομίζω ότι χρησιμοποιούνται... Ε, πολύ απάνθρωπες συνθήκες στη Λευκορωσία και νομίζω θα πρέπει να είμαστε σε θέση να τους βοηθήσουμε. Σε αυτή την περίπτωση είπα χτες ότι αμελητή θα πρέπει να ζητήσουμε από τον πρόεδρο Λουκασέγκο να εφαρμόσει μορατόριουμ στην θανατική Φανταστείτε να είσαστε μητέρα και ο γιος σας να έχει καταδικαστεί παρόλο ότι είναι αθώος και το γνωρίζουν όλοι και όμως αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή η οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί οποιαδήποτε σημεί και πολλές φορές δεν διατίθεται ούτε η σωρός του θανόντα. Αυτή είναι μια απάνθρωπη, απάνθρωπη κατάσταση στη χτεσινή συνάντηση. ε, μας ελέγχθη ότι θα αποσταλεί επιστολή επί του θέματος και ο κύριος Σούλς εξέφρασε αυτή την επιθυμία. Θεωρώ λοιπόν ότι εμείς ως υποεπιτροπή πρέπει να συντάξουμε αυτή την επιστολή ζητώντας μορατόριουμ για την εφαρμογή της θανατικής ποινής έτσι ώστε να ανασταλεί στο άμεσο μέλλον. Έτσι θα ενισχυθεί και το γόητρο της υποεπιτροπής μας. Αυτοί που μας επισκέφθηκαν χτες, οι επισκέπτες μας δεν θα κατανοήσουν αν δεν ζητήσουμε αυτό το μορατόριο. Δεν αρκεί το ότι το ανέφερε ο πρόεδρος μας, ο κύριος Σούλς. Θα πρέπει να συνταχθεί αυτή η επιστολή εξ ονόματός μας. Ευχαριστώ την κυρία Λόχ Μπίλερ για ό,τι έκανε το Δεκέμβριο, αλλά οι νέες πληροφορίες που έχουμε λάβει ε, σημαίνουν ότι θα πρέπει να παραβλέψουμε αυτή την δυνατότητα. Ας αποστείλουμε αυτή την επιστολή και έτσι θα ενισχυθεί και το γόητρο της Επιτροπής μας. Εντάξει. Υπάρχει συμφωνία προς το περιεχόμενο. Ξανακοίταξα το δελτίο τύπου του Μάρτιν Σούλτς και αναφέρει και εκείνος ε, το μορατόριουμ, όπως ε, το αναφέρει και η Λεδιάστον το Φεβρουάριο. Χρειάζεται όμως ε, και μεγαλύτερη υποστήριξη και αυτό θα γίνει αν όλοι οι αντιπρόεδροι και οι πρόεδρος στείλουμε ως Προεδρείο μια επιστολή στον πρόεδρο Λουκασέγκο και νομίζω ότι θα το προετοιμάσουμε καταλήλως. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Βάιντερε, ε, το εκτιμώ ιδιαίτερω. Σα ευχαριστούμε. Κυρία Γκόμας. Um, uh, um, um, ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόσφατα είχαμε τη δέκατη θλιβερή επέτειο από την ενέργεια λειτουργίας του Γκουαντάναμο, που δεν έχει κλείσει ακόμη. Παρά τις, υποχρεώσεις, υποσχέσεις του Πρόεδρου Ομπάμα. υπάρχουν κρατούμενοι στους οποίους δεν έχει απαγγελθεί η κατηγορία και ποτέ δεν θα τους απαγγελθεί η κατηγορία και ακόμη εκεί βρίσκονται. Χθε τρεις βουλευτές, ε, εγώ και η Αλίτ και η Τζιν Λάμπερτς οργανώσαμε μια συνεδρία με προβολή μιας ταινίας και με συμμετοχή κάποιων απελευθερωθέντων από το Γουαντάναμο και ο στόχος αυτών των ενεργειών είναι η απελευθέρωση αυτών των κρατουμένων που δεν τους έχει απαγγελθεί κατηγορία και βρίσκονται ακόμη στο Γκουαντάναμο. Συνδυάσαμε τις πρωτοβουλίες μας, εμείς οι τρεις, με προσπάθειες ε, κάποιου ο οποίος ε, ενδιαφέρεται για τα δικαιώματα των υπολείπων. Είναι κάποιος ο οποίος μπορούσε να μιλήσει και αγγλικά και τον θεωρούν ε, ως άτομο που μπορεί να έχει επιρροή με τρομοκρατικές τάσεις επειδή ακριβώς έχει αυτό το ρόλο ενώ αυτές οι κατηγορίες ποτέ δεν έχουν αποδειχθεί. Ονομάζεται ο Μάρ Σακύρ Μάλλον όχι. Σακίρ Μπέτς ονομάζεται. Αποφασίσαμε να στείλουμε μια επιστολή στον πρόεδρο Ομπάμα. Αυτό μπορεί να αποτελεί πρωτοβουλία κάποιων βουλευτών, όπως σας είπα ότι είμαστε εμείς οι τρεις. Αλλά εκ μέρους της υποεπιτροπής ενδέχεται να θέλετε να συνδυάσετε και τη συμμετοχή της Επιτροπής μας σε αυτή την πρωτοβουλία. Τώρα ο Πρόεδρος Ομπάμα θέλει να επανεκλεγεί. Και επίσης ο Πρόεδρος Ομπάμα έχει εγκρίνει ένα κανονισμό που επιτρέπει την απεριόριστη κράτηση αυτών των ατόμων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Γκόμες. Ο κύριος Φλίτ, ειδικό εκπρόσωπος, δεν ξέρω ακριβώς τον τίτλο του, τον έχει διορίσει ο πρόεδρος Ομπάμα, ήρθε πάντως πέρυσι στο Κοινοβούλιο και ζήτησε βοήθεια για να μπορούν και άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να δεχθούν περισσότερους κρατουμένους θα μπορούσαμε εκ μέρους της Επιτροπής Ντρουάν να στείλουμε μια επιστολή στον Πρόεδρο Ομπάμα σχετικά με αυτό που ζητάτε. Ο νέος νόμος για τη στρατιωτική πολιτική έχει αρκετές λεπτομέρειες που θα εμποδίσουν τον πρόεδρο Ομπάμα να κλείσει το Γκουαντάναμο. Θα μπορούσαμε όμως εμείς να εστιαστούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση και να το διευρύνουμε στην επιστολή μας. Κυρία Γκόμες. Θα ήθελα να ανακοινώσω στα μέλη της υποεπιτροπής μας ότι κάποιοι βουλευτές και εγώ μεταξύ αυτών έχουν δημοσιεύσει μία γραπτή δήλωση και θα θέλαμε να την προσυπογράψετε. Ε, κάτι το οποίο θα μεταβιβαστεί στον πρόεδρο Ομπάμα και στους συναδέλφους μας στο Αμερικανικό Κογκρέσο σχετικά με την ασυμβατότητα με το διεθνές δίκαιο ε, της ε, επιλεκτικής δολοφονίας με μη επανδρομένα οχήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Νομίζω τώρα μπορούμε να κλείσουμε το τμήμα των ανακοινώσεων της Προέδρου και περνάμε στην ανακοίνωση της Επιτροπής ε, παρουσίαση του νέου κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Μέσο για την Προαγωγή της Δημοκρατίας και των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Παγκοσμίω, κανονισμός ΕΜΔΑ. Και υπάρχουν και κάποια θέματα για τα υπόλοιπα προτινόμενα μέσα, όπως είναι το Μέσο Σταθερότητας, το Ευρωπαϊκό Μέσο Γυπνίασης και Εταιρικής Σχέσης και το Προενταξιακό Μέσο. Ε, καλωσορίζω και τον ε, Γκραφ Λάμστορφ, που είναι η συγητής του Κοινοβουλίου για τον κανονισμό για το μέσο ΕΜΔΑ και κάποιοι άλλοι εισηγητές ε, έχουν οριστεί για τα υπόλοιπα μέσα. Ο κύριος Κούκαν είναι εισηγητής για το μέσο γειτονία και τον βλέπω μεταξύ μας. Την Φρανσίσκα Μπράτνε, συνάδελφό μου που είναι ε, εισηγήτρια για το μέσο σταθερότητας, δεν τη βλέπω. Και ο κύριος Βίκινεν είναι εισηγητής για το προενταξιακό μέσο. Ούτε κι αυτός όμως είναι εδώ. Και έχουμε και ένα συνολικό εισηγητή, μια συνολική εισηγητή, την κυρία Γιαννάκου, για το πολιτές χρηματοδοτικό πλαίσιο. Οι συνάδελφοι από τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες φαντάζομαι ότι θα μεταφέρουν στους εισηγητές που δεν είναι παρόντες αυτά τα οποία θα συζητήσουμε τώρα εδώ. Θα ήθελα να δώσουμε καταρχήν το λόγο στον κύριο Κρίστιαν Σμιτ, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Δίνω το λόγο στην Επιτροπή. Ε, διορθώνω, είναι διευθυντής της, στη Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής για την Ανάπτυξη και είναι διευθυντής ε, για ανθρώπινη και κοινωνική ανάπτυξη. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας συγχαίρω για την εκλογή σας, συγχαίρω και τους αντιπροέδρους. Η Επιτροπή προσβλέπει στη συνεργασία μαζί σας και με τα άλλα μέλη του Προεδρείου. Πρώτη φορά εμφανίζομαι στην Επιτροπή σας και γι' αυτό θέλω να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα. Είμαι ο νέος Διευθυντής ε, για ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα. Είναι και οι συνάδελφοι εξ αριστερών μου που τους έχετε συναντήσει πολλές φορές, ενώ εγώ πρώτη φορά έρχομαι στην Επιτροπή σα. Αυτή η διεύθυνση ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνία των πολιτών, την την εκπαίδευση, την υγεία, πολλά θέματα που αφορούν την υποεπιτροπή σα. Χαίρομαι λοιπόν που βρίσκομαι εδώ και μπορώ να σα παρουσιάσω την πρόταση για τον κανονισμό από το 2014 μέχρι το 2020. Έχω και διαφάνειε, τι οποίε θα ήθελα να σα παρουσιάσω. Θα με βοηθήσει η Κριστίνα για να ε, προβάλλονται οι διαφάνειες. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή και είναι δύσκολο ε, να ε, έχει συγκεκριμένα αιτήματα η Επιτροπή. Όμω ε, είναι και κατάλληλη στιγμή για να έχουμε μεγαλύτερε επενδύσει στα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί όπω βλέπουμε σε ολόκληρο τον κόσμο είναι δυνατόν να επέλθουν αλλαγέ. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια κρίσιμη καμπή όσον αφορά τι αλλαγέ. Θα σα παρουσιάσω λοιπόν το θεματολόγιο τη αλλαγή, όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν αναφερθεί ω μία από τι βασικέ προτεραιότητε. Το ίδιο και για την αναθεώρηση τη πολιτική γειτονία. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή προτείνει και μία νέα προσέγγιση για την προσέγγιση του προϋπολογισμού όπου τίθενται όροι για τα ανθρώπινα δικαιώματα και παρά τις ε, δημοσιονομικές δυσκολίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστεύω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να υποβάλουμε τέτοια αιτήματα για αυξημένες επενδύσεις ε, στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τώρα, να σας πω δύο λόγια για το γενικότερο πλαίσιο, το σημείο 2. Το μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι το μοναδικό μέσο και τα χρήματα δεν είναι το παν τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως έχει πει και η Βερόνι Άστον, υπησέρχονται ε, και σε όλα τα άλλα μέσα, τους διαλόγους, διπλωματικά διαβήματα, πολιτικό, πολιτικούς διαλόγους και όλα τα άλλα μέσα που έχουν σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το μέσο για την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι το μόνο μέσο και δεν θα έπρεπε να είναι και το μόνο μέσο. Προς το παρόν είναι σχετικά μικρό, είναι μικρού μεγέθους σε σχέση με τα υπόλοιπα μέσα τα οποία παράλληλα υπάρχουν. Επομένως είναι πολύ σημαντικό η Επιτροπή να μην ασχολείται μόνο με τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα αυτό των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και στους άλλους τομείς και υπάρχει σαφώς συμπληρωματικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, με τη σταθερότητα και γι' αυτό πρέπει να συνδέσουμε αυτούς τους τομείς. Να σας πω δύο λόγια τώρα για τα αποτελέσματα και τα διδάγματα που έχουμε πάρει από την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο. Τώρα έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο πάνω από 800, πάνω από 800 έργα, εκ των οποίων ε, περίπου 100 είναι επιχειρησιακά και από τις προτάσεις μας βλέπετε ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες δράσεις. Θα επανέλθω όμως σε αυτές. Ε, τώρα το μέσο αυτό εφαρμόζεται σε 100 αντιπροσωπείες ε, τουλάχιστον. Είναι ένα μέσο το οποίο είναι παγκόσμιας εμβέλειας με διαφοροποιημένη προσέγγιση βέβαια παρόλα αυτά είναι ένα μέσο που απαιτεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πάνω από 100 χώρες. Πριν υποβάλουμε την πρότασή μας, ε, εξετάσαμε τις αξιολογήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Μία αξιολόγηση θα δημοσιευθεί σύντομα και εξετάζει την αποτελεσματικότητα του μέσου ε, αυτού και θα παρουσιαστεί αυτή η αξιολόγηση τον επόμενο μήνα σε μια ε, ευρεία ε, διοργάνωση. Θα ήθελα όμως να σας πω εγώ δύο βασικά πράγματα, ότι το μέσο αυτό επιτυχάνει αποτελέσματα, τοποθετώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση στο κέντρο της προσοχής. Αυτό είναι κάτι που το παραθέτω από την αξιολόγηση. Επίσης, από την αξιολόγηση για το μέσο αυτό, ένα άλλο έβριμα ε, ε, είναι ότι χρειάζονται αποφάσεις για να μπορέσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα να βγουν από το γκέτο στο οποίο συχνά το αφήνουμε. Το γκέτο είναι εδώ ο συνάδελφός μου εξ αριστερών και άλλα μέλη της μονάδας του που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή το μέσο το οποίο παίρνουμε από την αξιολόγηση είναι ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το μέσο αυτό θα μπορέσει να προσεγγίσει και τους άλλους τομείς. Θα επανέλθω όμως αυτό. Ε, λοιπόν, κλείνοντας αυτό το σημείο, βλέπουμε ότι πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη στρατηγική ευελιξία και περισσότερους πόρους. Πολλές φορές το έχετε ακούσει και πρέπει να το επαναλάβουμε. Ένα από τα τρία έργα επαρκούς ποιότητας μπορούν να χρηματοδοτηθούν με το τρέχον ε, χαρτοφυλάκιο που έχουμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερους πόρους. Όσον αφορά τώρα την ουσία του μέσου ΕΜΔΑ, όπω έχει δείξει η αξιολόγηση, είναι κάτι το οποίο λειτουργεί, επομένω δεν πρέπει να αλλάξουμε κάτι που λειτουργεί. Θέλουμε λοιπόν να το διατηρήσουμε. Υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που τα γνωρίζετε, απουσία συνένεση τρίτη χώρα και στην Επιτροπή σα δεν χρειάζεται να εξήγησω γιατί είναι ουσιαστικό αυτό το σημείο ευελιξία σε δύσκολες περιπτώσεις, πράγμα το οποίο το διαθέτει το μέσο ΕΜΔΑ και θέλουμε να το ενδυναμώσουμε και συμπληρωματικότητα με άλλα μέσα. Αποστολές παρατήρησης εκλογών είναι επίσης ένα σημαντικό τμήμα του τρέχοντος μέσου και θα παραμείνει ε, στην ε, πρόταση που υποβάλλουμε τώρα. Και τέλος, προτείνουμε να συνεχίσουμε να αποκλείουμε την άμεση χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων. Ευχαρίστως θα σας πω γιατί κάνουμε αυτή την πρόταση και θέλω να τονίσω ότι αυτό δεν συμπεριλαμβάνει την εργασία με πολιτικά ιδρύματα στην Ευρώπη που μπορούν να διευκολύνουν τον πλουραλισμό και την κατανόηση στις χώρες εταίρους. Αυτό μπορεί να συνεχίσει να είναι δυνατό στο μελλοντικό μέσο. Η άμεση χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων όμως θα εξαιρείται από την πρότασή μας. Ποιες καινοτομίες ε, παρουσιάζουμε στη νέα μας πρόταση. Οι στόχοι καθορίζονται σαφέστερα, όπως θα δείτε. Υπάρχει μεγαλύτερη υποστήριξη και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προωθούνται και υποστηρίζονται οι δημοκρατικές διαδικασίες, όπως θα δείτε στο σχέδιο κανονισμού. Δεύτερον, προσπαθήσαμε ε, να επικαιροποιήσουμε το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, ούτω ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις από το 2007, μεγαλύτερη έμφαση στα ε, κοινωνικά δικαιώματα, ε, στην ελευθερία της σκέψης, ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και ελευθερία του διαδικτύου. Δεν θέλω να διαφημίσω τα κοινωνικά δίκτυα, δεν χρειάζεται να το κάνω εγώ. Είναι μια σημαντική εξέλιξη και το δικό μας μέσο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα νέα μέσα που υπάρχουν διαθέσιμα. Τρίτον, προτείνουμε ε, ισχυρότερη στρατηγική εστίαση στις πιο δύσκολες χώρες, εκεί όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα διατρέχουν μεγαλύτερους κινδύνους. Θα επικεντρωθούμε περισσότερο λοιπόν εκεί. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια αύξηση των, ε, του ποσοστού εμπιστευτικών προγραμμάτων. Σας έδειξα προηγουμένως, 100 από τα 1.800 είναι εμπιστευτικά ε, και πρέπει να ενισχύσουμε αυτή την τάση στις ε, πιο δύσκολες περιπτώσεις. Όταν υπάρχει εμπιστευτικός χαρακτήρας θα πρέπει η Επιτροπή και η δική σας Επιτροπή ενδεχομένως να, βρει, να βρουν τον τρόπο άτυπης συνεννόησης για τέτοιου είδους εμπιστευτικά έργα. Εμείς ευχαρίστω θα διευκολύνουμε μια τέτοια συνεργασία. Τέλος, ε, εστιάζουμε στη δημοκρατία ως διαδικασία, όχι μόνο με αποστολές παρατήρησης εκλογών, αλλά παρακολουθούμε και τα όσα γίνονται μεταξύ εκλογών. Όπως είπα προηγουμένως, είναι σημαντικό να, βγούμε, να βγάλουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα από τον γκέτο. Δηλαδή να μην εξετάζουμε μόνο το μέσο για τη δημοκρασία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά να δούμε τι γίνεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και σε άλλα μέσα θα είναι τμήμα του πακέτου το οποίο υιοθετήθηκε μαζί με αυτό τον κανονισμό, το μέσο σταθερότητας, το μέσο γειτονίας και το μέσο προενταξιακής βοήθειας. Όλα αυτά τα μέσα συμπεριλαμβάνουν στους στόχους τους σαφέστατες διατυπώσεις ότι πρέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα να αποτελούν τμήμα των δραστηριοτήτων τους. Εδώ βλέπετε σε αυτό το slide την αντίστοιχη διατύπωση που υπάρχει στο μέσο για την προενταξιακή βοήθεια. Και προσπαθούμε να τα εκφράσουμε σαφέστερα στο νέο μέσο. Ε, εδώ βλέπετε το τρίτο σημείο που αφορά την ευελιξία. Αυτό το μέσο είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα, σε αυτό το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό της ευελιξίας. Πρέπει να διατηρήσουμε τη δυνατότητα άτυπων εταιρικών σχέσεων, να μπορούμε να συνεργαστούμε με εταίρους που δεν έχουν ε, νομικό καθεστώς, ε, δεν είναι νόμιμα, νόμιμες οργανώσεις ε, ε, και ε, στη χώρα τους και δεν υπάρχουν άλλα μέσα που να δίνουν αυτή τη δυνατότητα και σαφώς υπάρχουν, υπάρχει αιτιολόγηση ε, αυτό το μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα να έχει αυτή τη δυνατότητα ευελιξίας. Δεύτερον, θέλουμε να διατηρήσουμε τη δυνατότητα ανακατανομής κονδυλίων μέσα στα έργα και βλέπετε ότι υπάρχει και ένα προτινόμενο κατόφλι 100.000 ευρώ. Και τρίτον, έχουμε σχετική πείρα για ότι μικρά κονδύλια μέχρι 10.000 ευρώ για υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν αποτελέσει μεγάλη επιτυχία. Δυστυχώς, αλλά αυτή είναι η εμπειρία μας. Είναι πολλές οι περιπτώσεις ε, στις οποίες αξίζει τον κόπο να δίδονται τέτοιες ε, επιχορηγήσεις και προτείνουμε αυτή η επιτυχημένη εμπειρία να συνεχιστεί. Μια πολύ σημαντική καινοτομία είναι το προτινόμενο ποσό του προϋπολογισμού. Και ξεκινώ, επανέρχομαι σε αυτό με το οποίο ξεκίνησα, ότι λόγω της τρέχουσας κατάστασης αξίζει τον κόπο να επενδύσουμε στα ανθρώπινα δικαιώματα. Φαίνεται από τις γειτονικές μας περιοχές ότι είναι κάτι που αξίζει τον κόπο να το κάνουμε και είναι δυνατόν να έχει αποτελέσματα. Προτείνουμε λοιπόν μια αύξηση, ώστε να έχουμε ετήσιο προϋπολογισμό 225 εκατομμύρια ευρώ περίπου και ξέρουμε ότι είναι ποσό που μπορούμε να δαπανίσουμε. Δεύτερον, προτείνουμε ένα νέο μέσο για άμεση χορήγηση επιδοτήσεων στις πιο δύσκολες περιπτώσεις την ε, αρχή της διαφάνειας ε, και της δίκαιης επιλογής θα την κρατήσουμε, αλλά σε ορισμένε ε, περιπτώσεις, σε ορισμένες χώρες δεν είναι δυνατόν να διεξάγουμε, να κάνουμε προκήρυξη ε, υποβολής προτάσεων. Ε, σε ορισμένε περιπτώσεις λοιπόν, σε ορισμένες προφανείς περιπτώσεις έχουμε χώρες όπου μπορούμε να έχουμε άμεση ανάθεση. Αυτό ισχύει και στο μέσο σταθερότητα, όπου υπάρχει δυνατότητα μέχρι 2 εκατομμύρια ευρώ να δίδονται με άμεση ανάθεση. Υπάρχουν αρκετές απλουστεύσεις στον οριζόντιο κανονισμό κοινή εφαρμογή για όλα τα μέσα και μία από τις απλουστεύσεις είναι ότι αυτό το συγκεκριμένο μέσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν θα έχει δεσμεύσεις, θα είναι από δεσμευμένο και θέλουμε να είναι πραγματικά παγκόσμιο μέσο και να μπορούμε να έχουμε συνεργασία σε, παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή είναι η πρόταση της Επιτροπής για το μέσο ΕΜΔΑ. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω για τη Βερμανία που αναφέρατε νωρίτερα. Το μέσο χρησιμοποιείται ήδη Προτείνεται τώρα ένα νέο πακέτο από την Επιτροπή και αυξάνεται η παρέμβασή μας στη Βερμανία και θα χρησιμοποιήσουμε το μέσο για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα ως μέσο ε, για να υποκινήσουμε και άλλα πράγματα τα οποία κάνουμε, όπως είναι η αγροτική ανάπτυξη ε, και ο Επίτροπος Πίλμπαξ θα πάει στη Μιανμάρ ε, προσπαθώντας να εντείνει αυτή την προσπάθεια. Τώρα που ανοίγει η χώρα θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε το μέσο αυτό ως μέσο μόχλευσης και για όλους τους άλλους τομείς. Αυτά είχα να σας παρουσιάσω και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Με χαρά θα συζητήσουμε την πρόταση αυτή μαζί σας και ελπίζουμε ότι θα τύχει ευνοϊκή υποδοχή από εσά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σμιτ. Έχω δύο ερωτήσεις πριν ε, ξεκινήσει η συζήτηση. Πρώτα απ' όλα μπορείτε να μας δώσετε την παρουσίαση αυτή για να την δώσουμε στους συναδέλφους και δεύτερον δεν κατάλαβα πώς συνεργάζεστε με την υπηρεσία εξωτερικών υποθέσεων, π.χ. με την Διεύθυνση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Εξηγήστε μας αυτό το κομμάτι μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Νομίζω κ. Λάμσδορφ είναι ο εισηγητής. Έχετε λοιπόν το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Κομισιόν για την παρουσίαση του μέσου αυτού. Πράγματι το μέσο αυτό είναι κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για ευρωπαϊκές αξίες και έχει μεγάλη σημασία αυτό για την παγκόσμια υπεράσπιση τους. Και βεβαίως καλό είναι να το αξιολογούμε και να προτείνουμε και καινοτομίες Έχω και εγώ το ίδιο ερώτημα με εσά, κυρία Πρόεδρε. Πώς έχει η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, γιατί βεβαίως ε, πρέπει να μας πει κάτι κομισιόν για τη νέα κατάσταση. Σημαντικό νομίζω αυτό. Επίσης, σωστό είναι αυτό που ακούστηκε, ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο κλειδί Είδαμε πως υπάρχουν ελλείψεις. Ειδικά όσον αφορά την πρόθεση της δημοκρατίας στο μέσο αυτό και στην γειτονιά μας και στη Βόρεια Αφρική. Μας εξέπληξαν εκεί οι εξελίξεις και το πρώτο ερώτημα που σχετίζεται άμεσα με αυτό, όταν μιλάμε για δημοκρατία και πρόθεση της δημοκρατίας, η Κομισιόν θα ήθελε να σταματήσει την άμεση στήριξη πολιτικών κομμάτων από αυτό το μέσο. Εδώ πέρα έχει σκεφτεί η Κομισιόν ε, πώς μπορούμε αυτό να το δούμε συμπληρωματικά από ένα μέσο ε, τέλος πάντων ε, ταμείο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Δημοκρατίας τι σκέψεις κάνετε σχετικά. Δεύτερο ερώτημα. Τον επόμενο μήνα βεβαίως ε, θα ήθελα να ακούσω τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Ε, εγώ δεν σας είχα για παιδιά του γκέτο, εν πάση περιπτώσει. Ε, δεν ξέρω ο κύριος Νίλο θεωρείται ότι ζει στο γκέτο, αλλά αν μπορούμε να βγάλουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα από το γκέτο, Βεβαίω να βοηθήσουμε ω κοινοβουλίο. Αλλά κάποιες ερωτήσει Είπατε πως μία από τις δυνάμεις ε, του μέσου αυτού είναι η συμπληρωματικότητά του με τα άλλα μέσα, αλλά μετά στο τέλος παρουσιάζεται μία νέα πιθανότητα δυνατότητα άμεσης χρηματοδότησης και είπατε πως κατά βάση είναι παρόμοιο με αυτό το οποίο υπάρχει στο μέσο σταθερότητας. Αυτές οι άμεσες χρηματοδοτήσεις μέχρι 2 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ πέρα τίθεται το ερώτημα γιατί υπάρχει αυτό σε δύο μέσα. Είναι αναγκαία αυτή η δουλειά να γίνει δύο φορές. Το δεύτερο ερώτημα που έχω είναι αυτό της ε, ε των ε, κονδυλίων γιατί μου παραπονιούνται συνεχώς η ΜΚΟ το πόσο δύσκολο είναι η διαδικασία αίτησης και νομίζω υπήρχε και η ιδέα από την Πολωνική Προεδρία να υπάρξει ένα πιο ευέλικτο μέσο και λέτε πως θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό πλαίσιο για την εφαρμογή. Συγκεκριμένα τι προγραμματίζετε εδώ πέρα. Ξέρω βέβαια πως δεν είναι αυτή δική σας ε, αρμοδιότητα, απλά θα ήθελα να ακούσω πώς, τι άποψη έχετε. Τελευταίο τώρα και θα ήθελα να ακούσω κάτι παραπάνω όσον αφορά την ουσία γιατί στην ανάλυση συμφωνούμε εδώ και χρόνια. Είναι η προσέγγιση του εκλογικού κύκλου στην πρόθεση της δημοκρατίας. Ε, είχα πάει και εγώ σε πολλές ε, προστολές παρατήρησης εκλογών. Ξέρω πώς λειτουργεί αυτό, αλλά ξέρω πόσο δύσκολο είναι να υπάρξει μια γενικότερη στήριξη της ε, δημοκρατίας ανεξαρτήτως από τον κύκλο των εκλογών. Δεν υπάρχει καλή αλληλεπίδραση. Εσείς είπατε πως θέλετε μια δημοκρατία ως διαδικασία για ολόκληρο τον δημοκρατικό κύκλο. Τι ακριβώς σκέφτεστε εδώ. Κατά λοιπά χαίρομαι για την ε, συνεργασία μαζί σας και με τον κύριο Λαμό για τους πολύ σημαντικούς αυτούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Λάμσδορφ, αν συμφωνείτε κύριε Σμιτ, νομίζω α, ακούσουμε και άλλες ερωτήσεις και μετά. Κυρία για έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, συγχαρητήρια για την εκλογή σας. για τα θέματα αυτά. Έχω κάποιες ερωτήσεις και από τη σκοπιά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και του υπόλοιπη δουλειά μου εδώ πέρα, δηλαδή από τη γεωργική πολιτική και τις διμερείς συμφωνίες που κλείνουμε και το πώς μπορούμε να λάβουμε υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα ή τα δικαιώματα των εργαζομένων επιτόπου στις χώρες αυτές σε ποιο βαθμό μπορούμε να υποστηρίξουμε κάτι τέτοιο με αυτό το μέσο. Δηλαδή, την ανάπτυξη της υπαίθρου, κάτι το οποίο κατά την άποψή μου θα μπορούσε να αποτελέσει μια εξαιρετική βάση αναπτυξιακής βοήθειας και ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατά το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, γι' αυτό το αναφέρω, γιατί το ίδιο ακριβώς αναφέρθηκε από την Δανική Προεδρία χτες ε, στην Επιτροπή Γεωργίας και ήταν συναρπαστικό να δούμε αυτή την πτυχή στις εμπορικές ε, συμφωνίες. Και το ερώτημά μου είναι, μια που μιλάτε για μόχλευση εδώ πέρα, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και αν ναι, υπό ποια μορφή, πώς μπορεί να διαμορφωθεί η ροή των κονδυλίων. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε και από τις δύο πλευρές και κατόπιν από την Σκοπιά της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πώς μπορούν οι μικρές κοινότητες η οικογένειες ή ένας αριθμός οικογενειών να ενωθούν για να υπάρχει αυτή η προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Γιατί το πρόγραμμα leader ε, στη γεωργική πολιτική έχει μια τέτοια ακριβώς προσέγγιση. Ε, Δήμοι, ενώσεις, ε, συνεταιρισμοί πρέπει να έχουν ιδέα για το τι θέλουν να ζητήσουν από τις Βρυξέλλες και μετά ζητάνε λεφτά. Ξέρετε κυρία Λοχμπίλερ πως αυτό λειτουργεί καλά στη Γερμανία. Εγώ δεν βλέπω λοιπόν εδώ πέρα το πώς θα μπορούσαμε αυτό να το συνδέσουμε με τα δύο αυτά επίπεδα. Σας ευχαριστώ. Κυρία Βαϊντέρε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Έχω και εγώ ένα ερώτημα που σχετίζεται με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Λάμσδορ. Πρακτικό. Πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός για την άμεση χρηματοδότηση. γιατί ο κύριος Λάμζορφ είπε πως οι ΜΚΟ έχουν δυσκολίες. Ε, μπορείτε λοιπόν, σας παρακαλώ κύριε Σμιτ, να μας εξηγήσετε πώς λειτουργεί. Πώς γίνονται οι αιτήσει, πρακτικά πώς γίνεται η διαδικασία. Ευχαριστώ, Ρίτσαρτ Χάουιτ. Πρώτα απ' όλα, Πρέπει να θυμόμαστε πως ε, την προηγούμενη φορά που είχαμε πρόταση για εξωτερικά μέσα ήταν ε, πριν από πέντε χρόνια και είχε προτείνει τότε η Επίτροπος να καταργηθεί τελείως το μέσο αυτό. Ε, τώρα έχουμε μια πιο επικοδομητική θέση θα έλεγα. Μιλάμε για ενίσχυση του μέσου αυτού. Θα ήθελα να καλωσορίσω και εγώ τον κύριο Σμιτ Ελπίζω να έρχεστε τακτικά στην Επιτροπή μας και να συνεργαστούμε και να συνεργαστείτε με την υπηρεσία εξωτερικής ε, δράσης. Όλοι προσπαθούμε να μάθουμε τις νέες αυτές σχέσεις. Είμαι σίγουρος πως αυτή είναι και η δική σας ε, πρόθεση. Εμείς στηρίζουμε τις αρχές της στήριξης των υποστηρικτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, εντάξει, ήταν λίγο ηρωνικός λέγοντας πως δυστυχώς έχει μεγάλη επιτυχία το μέσο, αλλά πρέπει νομίζω να επενέσουμε τις αντιπροσωπείες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν παρεμβαίνουν, όταν απειλούνται οι υπερασφιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι κάτι το οποίο εκτιμάμε στην υποεπιτροπή μας, οπότε είναι ένα ευχάριστο πρόβλημα βεβαίως, αν και οι άνθρωποι, οι ενδιαφερόμενοι είναι απελπισμένοι. και Βεβαίω ε, θα έπρεπε να δούμε αν μπορούμε να έχουμε κάποιο συστηματικό μηχανισμό για τους υπερασπιστές εκείνους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που ε, αναγκάζονται να ζητήσουν να βρουν καταφύγιο στην Ευρώπη. Για το ζήτημα της αποδέσμευσης αυτού του ζητήματος πράγματι ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχετε δίκιο αν και νομίζω έχουν δίκιο οι συνάδελφοι με τις ερωτήσεις για τα άμεσες χρηματοδοτήσεις πρέπει να υπάρχει κάποιος έλεγχος βεβαίως πολλοί συνάδελφοι ε, αντιλαμβάνονται πως νομίζω το, το χειρότερο είναι να το συζητήσουν στην Επιτροπή προϋπολογισμού και να αρχίσουν να μιλάνε για προσφορές και τέτοια πράγματα και να μην καταλαβαίνουν τι θα πει κρίση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τούτου ρεχθέντο. Απογοητεύτηκα για το ότι δεν μιλήσατε για τον δομημένο διάλογο της Επιτροπής μας ε, με την Κομισιόν που έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια σε σχέση ακριβώς με το μέσο αυτό δεν είναι τέλειες οι συναντήσεις ε, όσον αφορά τη λογοδοσία, αλλά είχαμε πολύ επικοδομητικές ε, συναντήσεις, συζητήθηκαν και κλεισμένων των θυρών ε, τα εμπιστευτικά ζητήματα, με τρόπο που ελπίζω να βοήθησε και τους εμπλεκομένους, τους εξωματούχους και τους βουλευτές. Και οπωσδήποτε έχει τεθεί αυτό το ζήτημα και στην Ολομέλεια με τον Επίτροπο Φούιλε και την κυρία Άστον Οπότε πρέπει να, να τα λέτε αυτά, μην σας τα υπενθυμίζουμε εμείς. Πρέπει να πείτε πως ε, είναι σωστός αυτός ο δομημένος διάλογος. Γιατί είναι νομίζω μέρος αντιμετώπισης του προβλήματος της εμπιστευτικότητας και της λογοδοσίας. Όσον αφορά... Δεν βγάζω τα γραμματά μου. Α, ναι, αναφέρατε κάτι το οποίο είναι νομίζω σημαντικό για την συμφωνία με το Συμβούλιο και την Κομισιόν για τον έλεγχο από το Κοινοβούλιο μετά το 2014. Μα κοιτάξτε, μην τα λέμε εμείς, πείτε τα εσείς, θα έχουμε συναπόφαση στα έγγραφα στρατηγικής ως Κοινοβούλιο και θα μπορούμε να επηρεάσουμε τις προτεραιότητες μετά το 2014. Είναι περίεργο το ότι δεν είναι αυτό στην ε, παρουσίασή σας. Ο ε, δε κύριος Λάμστορφ δεν είπε τίποτα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία και μου φάνηκε περίεργο. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, το συζητάμε εντός Κοινοβουλίου, προσπαθεί να συμβιβάσει τις απόψεις ε, όταν μιλάμε π.χ. για χρηματοδότηση κομμάτων, πότε είναι ένα κόμμα κόμμα, πότε είναι κίνημα, πότε είναι ε, ένα εθνικό κίνημα. Πηγαίνετε στην πλατεία τα χρήρη και πείτε μου πώς κάνετε αυτές τις διακρίσεις. Δεν και εσείς δεν το ξέρετε και εγώ δεν το ξέρω. Αλλά εάν πρόκειται να συνεισφέρουμε στην Αραβική Άνοιξη πρέπει να βοηθήσουμε την αντιπολίτευση. Το ερώτημα είναι πώς το κάνουμε. Ίσως το Ταμείο για τη Δημοκρατία είναι ένα τέτοιο στοιχείο. Και η κυρία Γκόμες νομίζω ε, είναι υποστηρικτής. Αλλά μην το αγνοείτε, γίνεται μια συζήτηση. Να είμαστε όριμοι. Τρία ακόμα σημεία. Στον θεματικό κατάλογο, το μέσο, την τελευταία φορά που συζητήσαμε, ε, για επιχειρήσεις και ανθρώπινα δικαιώματα. Μπορείτε να μας πείτε αν εξακολουθεί να υπάρχει ως θεματική προτεραιότητα και οπωσδήποτε τα ζητήματα ΛΟΑΤ είναι πολύ ευαίσθητα σε πολλές χώρες και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Ε, αναφέρονται ε, ως θεματικό ζήτημα στην πρόταση. Και τέλος, αναφέρεται κάποια σημαντικά πράγματα για την ενσωμάτωση πολιτικών Όλοι είναι υπέρ. Η τελευταία δε προσπάθεια δεν ήταν ενσωμάτωση αυτού του μέσου, ήταν απόπειρα καταστροφής του. Γι' αυτό το στηρίξαμε. Εμείς δεν θέλουμε όμω να είναι χωριστά. Το στηρίζουμε πλήρω. γι' αυτό σα καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για αυτό το οποίο έκανε οι συνάδελφοί σα ε, σε σχέση με τα άλλα μέσα. που ήταν εξαιρετικά πράγματα. Αλλά το ΕΜΔΑ είναι μικρό ποσό σε σύγκριση με τα υπόλοιπα εξωτερικά μέσα. Αυτό το οποίο χρειάζεστε είναι όχι μόνο οι αρχές της ενσωμάτωσης στην πολιτική, αλλά μηχανισμοί για να λέμε πρώτα απ' όλα γιατί όχι το γεωγραφικό μέσο και αν υπάρχει κάποιος λόγος να είναι το ΕΜΔΑΒ, εντάξει, καλώς. Αλλά δεν το αναφέρατε στην παρουσίασή σας και πραγματικά α, με ενδιαφέρει είναι το πώς εφαρμόζονται αυτά τα οποία είπατε. γιατί λέμε π.χ. μικρές επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις πρώτα. Πώς θα πούμε πρώτα ενσωμάτωση στην πολιτική ε, είναι κάπως σκληρές οι ερωτήσεις μου, αλλά έχουν στόχο να βελτιωθούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Γκόμες. Ε, ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ε, ευχαριστήσω τον κύριο Σμιτ για την παρουσίασή του Είχαμε ε, μία πολύ καλή ανταλλαγή απόψε τα τελευταία χρόνια με πολύ χρήσιμες πληροφορίες, ιδιαίτερα ως προς τα σχέδια που πρέπει να υπόκεινται σε ε, σχήματα εμπιστευτικού χαρακτήρα. Θα ήθελα, με βάση αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, να ρωτήσω το εξής. Και με βάση αυτά μόλις είπε ο Ρίτσαρντ Χάουιτ, θα ήθελα να πω γιατί δεν υπάρχει νομική βάση για κατεξουσιοδότηση πράξη, γιατί δεν εφαρμόζεται η νομική βάση για τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξης ε, στο ΕΜΤΑ. Επίσης, Θα ήθελα να ρωτήσω πώς βρίσκεται τρόπο συνεργασίας με το κοινοβούλιο. Έτσι, ώστε να χρησιμοποιηθούν και άλλα μέσα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την πρόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως το EMP και το DCI γιατί δεν τα χρησιμοποιείτε σε χώρες όπου ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, πολλές αντιφάσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποτίθεται ότι προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία και τα διάφορα συμφέροντα ιδιαίτερα ως προς την ε, αναπτυξιακή βιομηχανία, η οποία συνεχίζει την πορεία της σαν να μην έτρεχε τίποτα. Σκέφτομαι, έχω κατά την Αιθιοπία, η οποία λαμβάνει πολλά κοινοτικά κονδύλια και είναι και εκτός ε, μέσου που ελέγχει το Κοινοβούλιο, διότι δεν εντάσσεται ούτε καν στο DCI και, το DCI, και δεν ελέγχεται από το Κοινοβούλιο. Πώς θα ελέγξουμε λοιπόν αυτά τα κονδύλια τα οποία χορηγούνται σε μια χώρα όπως την Αιθιοπία που υποτίθεται ότι θα πρέπει να υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και επιτρέπουμε σε αυτούς που τα παραβιάζουν να δρούν ανενόχλητα και να κινούνται ανενόχλητα. Επίσης, σε σχέση με αυτά που είπε ο Ρίτσαρντ, Πιστεύω ότι θα ε, πρέπει να ε, προωθούμε αυτό το μέσο υπέρ της δημοκρατίας και δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να χρηματοδοτούμε και κόμματα μέσω του ΕΜΤΑ. Όμως, δεν ξέρω κατά πόσο εμείς θα κάνουμε τη διαφορά στις χώρες όπου υπάρχει μία αναδυόμενη δημοκρατία και όπου προσπαθούν ε, να, σε χώρες προσπαθούν να απαλλαγούν από μία ε, δικτατορία. Και νομίζω ότι το μέσο γειτονία της ε, προσνότων χώρες θα μπορούσε να βοηθήσει. Ας πάρουμε τη Λιβύη, όπου δεν υπήρχαν πολιτικά κόμματα καν. Πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε μια δημοκρατική διαδικασία με τις επικείμενες εκλογές όπου ε, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε στη δημιουργία πολιτικών κομμάτων. Εδώ θα πρέπει να προωθήσουμε τη δημοκρατία. Δηλαδή να υπάρχει ένα συνενετικό πλαίσιο για την εφαρμογή αυτού του μέσου. δηλαδή εκεί όπου πραγματικά υπάρχει δημοκρατική ατζέντα και δυνατότητα δημιουργίας πολιτικών κομμάτων. Θα ήθελα τα σχόλιά σας και επ' αυτού. Και μου κάνει εντύπωση γιατί αντί να έχουμε την, τον έλεγχο αυτού του μέσου, μέσου υπέρ της δημοκρατίας μέσα στα πλαίσια αυτού του δημοκρατικού φάσματος, επιτρέπουμε τον εθνικό έλεγχο, με την εθνική δηλαδή ε, ατζέντα, μέσω εθνικής ατζέντας. Επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς μπορούμε μέσω έμβα με μπερδεύει πολλές φορές αυτό το ακρονίμιο πώς μπορεί εν πάση περιπτώσει να χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπίσουμε τη διαφορά η οποία σχετίζεται πολλές φορές άμεσα με την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δηλαδή να το δούμε υπό αυτή την οπτική γωνία, όπως είπε και ο Ρίτσαρτ, δηλαδή των επιχειρήσεων, του επιχειρήν και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ε, παραβίασής τους, που θα πρέπει να μας απασχολήσει στο εξή. Ο κύριο Σταβάρες. Ευχαριστώ. Θα ήθελα εντάχει να ρωτήσω το εξή. Θα ήθελα να μου δώσετε ένα απτό παράδειγμα του πώς λειτουργεί αυτό το πλαίσιο σε μια χώρα τη στιγμή που ε, γίνονται διαγωνισμοί πώς έχουν τα ε, σχέδια εμπιστευτικού χαρακτήρα. Ιδιαίτερα για τη χορήγηση ε, κονδυλίων. How are the mechanics of the, of, of particular... Πώς λειτουργούν λοιπόν αυτά τα πλαίσια χορήγησης ε, κονδυλίων, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν ε, διάφορες, όταν υπάρχει φήμωση του τύπου, δηλαδή ε, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ε, μία εφημερίδα και πώς μπορούν να κινηθούν οι άνθρωποι μέσω blog ή κοινωνικών network. Πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε με λίγα λόγια έτσι ώστε να χορηγηθούν αυτά τα κονδύλια και να μπορούμε να ελέγξουμε και πώς δαπανώνται. Εάν δεν χρηματοδοτούμε πολιτικά κόμματα, πώς είσαστε σίγουροι ότι τελικά δεν χρηματοδοτούνται, παρόλο που δεν το επιθυμούν. Επίσης, πώς ξέρουμε τι λειτουργεί και τι όχι. Μπορούμε να έχουμε και κλεισμένων των θυρών συναντήσεις με τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Δηλαδή να συνομιλούμε με τους ανθρώπους που την χάνουν χρηματοδότησης. Να μας δώσετε ένα απτό παράδειγμα με βάση την ε, πείρα σας για να δούμε κατά πόσο έμπρακτα λειτουργεί κάτι τέτοιο σε αυτές τις χώρες. Ο κύριος Μακμίλαν Σκότ, ο αντιπρόεδρος μας, ε, προήγε αυτό το μέσο και είχε συνεισφέρει και στην σύστασή του. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Να σας συγχαρώ καταρχήν για την επανεκλογή σας, καθώς και τους αντιπροέδρους και συντονιστές, οι οποίοι εξελέγησαν ή επανεξελέγησαν σήμερα. Έχω δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για τη δραστηριότητα αυτής της Επιτροπής. Και η επιλογή η εισηγητρίας για το ΕΜΔΑ είναι πολύ καλή. Τώρα θα δούμε πώς θα οριστούν και οι σκιώδεις. Θα ήθελα να συγχαρώ και τα νέα μέλη, δηλαδή τον Λορέντσο, ε, το προσωπικό μας, το οποίο ήρθε από άλλες επιτροπές. Και ο Ραλφ Τίμανς ε, μου είπε «Α, να ξαναβλεπόμαστε μέσα στα, μέσα στα πλαίσια αυτού του κανονισμού». Έχουμε δοθεί και στο ε, παρελθόν. Η κυρία Φλότρ ήταν ε, συνεισηγήτρια στο παρελθόν για την έκθεση αυτή. Τώρα έχουμε ένα καλά οργανωμένο πρόγραμμα και για τους ψηφοφόρους μας, γιατί το ε, πρόσφατο ευρωβαρόμετρο που δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα ε, δείχνει ότι το κοινό θέλει να κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή είναι, αυτό είναι ένα από τα δεδομένα ως προς τις ε, φιλοδοξίες μας και τις φιλοδοξίες του κοινού. Ως προς το έμβα, ακολουθήσαμε τον ίδιο κύκλο, την ίδια πορεία γιατί πριν, α, πριν να πέσει το τείχος του Βερολίνου είχε εκφραστεί ανάγκη ενός εξειδικευμένου μηχανισμού για να προωθήσουμε τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπήρχαν μικρά προγράμματα, αλλά τίποτα το συντονισμένο. Και μετά είχαμε μεγαλύτερη όρεξη και διάθεση, μετά την πτώση του τείχους να φτάσουμε σε κάτι το σημαντικότερο χρειάστηκαν τουλάχιστον δύο ή μερικά χρόνια μέχρι το 1999 έτσι ώστε να προσθεθεί αυτό το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως ε, πλήρες ε, ε, πρόγραμμα. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει διαφορετική προσέγγιση με τη ΣΥΠΑ, διότι εμείς θεωρούμε το τα ανθρώπινα δικαιώματα σαν αναπόσπαστο μέρος της δραστηριότητάς μας, με βάση και τα δεδομένα του Συμβουλίου. Γι' αυτό χαίρομαι που προτείνεται αύξηση του προϋπολογισμού, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει εξέλιξη στον αραβικό κόσμο και αυτή η ανελικτική πορεία δεν έχει ολοκληρωθεί, όπως είπε και ο κύριος Χάουιτ. Και ο κύριος Λάμστορφ ε, ε, είπε ότι το, το θέμα αυτής της ε, πρικοδότησης δεν αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του προγράμματός μας. Λυπάμαι που δεν άκουσα τις προηγούμενες ε, παρεμβάσεις, αλλά η μικροχρηματοδοτήση μέχρι 10.000 ευρώ ήταν ε, πολύ επιτυχημένες. Αλλά είδαμε ότι μόνο πέντε ακολούθησαν αυτή τη διαδικασία ε, πρικοδότησης μέσω ΕΜΔΑ. Όταν λοιπόν μιλάμε για αυτή την πρικοδότηση θα πρέπει να έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα γιατί βλέπω ότι το έμδα γίνεται ένα ολένα και διονγκούμενος γραφειοκρατικός μηχανισμός. Δηλαδή μιλάμε για αναπτυξιακή πορεία και όχι για πολιτική καθαρά. Πολιτική ανελικτική πορεία. Και πολλές φορές στην Κομισιόν και στο Κοινοβούλιο ακολουθούμε μια διαδικασία πραγματογνωμοσύνης. Βεβαίως υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία από ό,τι στο παρελθόν, αλλά δεν διαθέτουμε ένα μηχανισμό ο οποίος να μην αμφισβητείται. Οι ΙΠΑ ακολουθούν μια διαδικασία χρηματοδότησης η οποία είναι απαράλλακτη και η οποία μπορεί να χρηματοδοτήσει και πολιτικά κινήματα ή κόμματα. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ένα βήμα προς τα πίσω και να κοιτάξουμε και προς αναταλάς. Να δούμε δηλαδή κατά πόσο εμείς διαθέτουμε ένα μηχανισμό υπέρ της δημοκρατίας όπως θα θέλαμε. Γιατί πολλοί προσμένουν περισσότερα από μας και μας θεωρούν πλέον ένα γραφειοκρατικό μηχανισμό. Δεν μιλάμε μόνο για ενίσχυση του ΕΜΔΑ. Χαιρόμαστε για τη συνεργασία μεταξύ Κομισιών και Κοινοβουλίου. Θα πρέπει όμως να αρχίσω μια σοβαρή συζήτηση για τον μηχανισμό πρικοδότησης υπέρ της δημοκρατίας. Και εγώ θα ήθελα να υποβάλω μια ερώτηση. Ήρθα σε επαφή με εκπροσώπους της κοινωνίας των ε, πολιτών, οι οποίοι φοβούνται ότι η Επιτροπή θα μειώσει τις χρηματοδοτήσεις ε, ως προς εσωτερικά ε, ζητήματα, εσωτερικά ζητήματα για τις ε, χώρες αυτές. Θα γίνει αυτό πράγματι. Και θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο θα μπορέσετε, θα μπορέσετε να υποστηρίξετε και τους αυτόχθονες ε, ο κύριος ε, Τίμανς ε, δεν μπόρεσε να είναι εδώ εξ αρχής. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο στον κύριο Σμιτ καταρχήν και στη συνέχεια στον κύριο Τίμανς. Έχετε το λόγο κύριε Σμιτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και όλα τα μέλη της Επιτροπής για το ενδιαφέρον και για την υποστήριξή σας. Δεν θα έχω το χρόνο να απαντήσω λεπτομερώς σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά τις έχω σημειώσει και θα ζητήσω και από τον Πατχής να λάβει το λόγο. Ε, ρωτήσατε και για τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τώρα που είναι εδώ και ο Ρόλφ μπορώ να πω ότι είναι εξαιρετικές οι σχέσεις μας. Το απόγευμα ολόκληρη η διεύθυνσή μας ε, θα συναντηθεί με την ομάδα της κυρίας Μαρινάκη και θα συζητήσουμε τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πυρηνικής ασφάλειας, μη διάδοση των όπλων έχουμε καλές λειτουργικές σχέσεις, ειδικά στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ε, έχει αποδειχθεί, υπάρχει μια πρόκληση και πρέπει να δούμε πώς αυτό το μέσο μπορεί να μπει μέσα στη γενικότερη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή η επισκόπηση των δικαιω... του θέματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς αυτό προσπαθεί να δει, κατά πόσο είναι συνεπής η πολιτική μας, κατά πόσο εφαρμόζουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά κλπ. Το μέσο υπάρχει, αλλά το μέσο ε, ε, είναι και πέραν αυτής της, υπάρχει και πέραν αυτής της ε, ε, επισκόπησης. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η πρότασή μας εγκρίθηκε στην Επιτροπή πριν οριστικοποιηθεί ε, η εξέταση, η επισκόπηση αυτή. Υπάρχουν όμως ε, σαφώς κάποια σημεία τα οποία είναι κοινά και μπορούμε να τα βρούμε και στα δύο. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, αναπτύσσει έγγραφα στρατηγικής αναχώρα, τα συζητάει με τις αντιπροσωπείες και το ίδιο είναι το προσωπικό που χειρίζεται και τα θέματα του μέσου. Τα συζητούν με τα κράτη-μέλη και έτσι προκύπτει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε κάθε δεδομένη χώρα. Και βέβαια θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις στρατηγικές ε, για να εντοπίσουμε τις ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε κάθε συγκεκριμένη χώρα όταν χρησιμοποιούμε το μέσο. Άρα λοιπόν όχι απλώς έχουμε καλές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, αλλά ξεκινάμε μια ενισχυμένη συνεργασία με αυτά τα έγγραφα πολιτικής και με τις δράσεις μας επιτόπου προς τον εισηγητή θέλω να πω ότι προσβλέπουμε σε μια καλή συνεργασία μαζί σας και με ρωτήσατε συγκεκριμένα για τα πολιτικά κόμματα, για το τι και πώς. Στην πρότασή μας λέμε ότι δεν θα συνεργαζόμαστε απευθείας με πολιτικά κόμματα, αλλά όταν θέσατε το θέμα της Αιγύπτου, παραδείγματος χάρη, μπορώ να πω ότι μπορούμε να προσφέρουμε ευκαιρίες για δημιουργία προϋποθέσεων σε όλα τα πολιτικά κόμματα που πρέπει να ενισχυθούν. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τους κανόνες της πολυφωνίας, να βοηθήσουμε στο πώς λειτουργεί και οργανώνεται ένα κοινοβούλιο κλπ. Αυτά είμαστε έτοιμοι να τα κάνουμε εφόσον ε, επιλέξουμε αυτόν με τον οποίο θα συνεργαστούμε για το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και για τα κονδύλια που διαθέτουμε, η θέση της Επιτροπής είναι ότι θεωρούμε ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία ε, για τις χρηματοδοτήσεις αυτές. Ξέρω ότι διαφέρουν οι απόψεις των κρατών μελών επί του θέματος. Στην Επιτροπή σας νομίζω μπορώ να πω ότι θα ήταν κρίμα να δημιουργήσουμε αυτή τη δυνατότητα παροχή κονδυλίων και χωρί να προσθέσουμε κονδύλια να αφαιρέσουμε χρήματα από το μέσο για να χρηματοδοτήσουμε αυτά τα άλλα κονδύλια. Όταν ήδη υπάρχει ένα μέσο που έχει ανεπαρκεί πόρους. Σαφώς υπάρχει λοιπόν προστιθέμενη αξία διότι αυτά τα κονδύλια που δίδονται για τη δημοκρατία δείχνουν ότι η Ευρώπη θέλει να είναι πιο ενεργός παίκτη σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά θα ήταν κρίμα αν μειώνουμε το μέσο ε, διαθέτοντας κονδύλια από αυτό. Σχετικά με την ευελιξία και το τι θα κάνουμε θα δώσω το λόγο στον Πατρίς να απαντήσει. Λίγο πολύ ακολουθούμε αυτό το οποίο γίνεται στο μέσο για τη σταθερότητα. Ζητούμε από τους εταίρους μας ε, πληροφορίες και ε, συνεχίζουμε με διαπραγματεύσεις με τους πιθανούς αποδέκτες μέχρι ότου καταλήξουμε σε παροχή χρηματοδότησης. Ο κ. Σταβάρης μου ζήτησε ένα παράδειγμα του πώς θα λειτουργούσε κάτι τέτοιο στην πράξη. Να σας πω στη Συρία τι γίνεται συγκεκριμένα. Φαντάζομαι ότι θα συμφωνείτε ότι η Συρία δεν είναι χώρα που μπορεί υπό τις τρέχουσες συνθήκες να κάνει κανείς προκήρυξη διαγωνισμού αποφασίσαμε ότι το θέμα ε, της λογοκρισίας στο διαδίκτυο είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή, ώστε να μπορούν να βγαίνουν οι φωτογραφίες, να έχουμε εικόνες από το τι συμβαίνει στη Συρία. Επομένως προσπαθήσαμε ε, να διαπραγματευτούμε με μη κυβερνητικές οργανώσεις εκεί για να τις υποστηρίξουμε και να μπορέσουμε να έχουμε εικόνες από την τρέχουσα κατάσταση στη Συρία. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα του πώς ε, λειτουργούν στην πράξη αυτό, ε, λειτουργεί στην πράξη αυτό το σύστημα με ευελιξία. Ο εισηγητής με ρώτησε ε, και για τη σχέση μας με τις επιστολές, αποστολές παρακολούθησης εκλογών. Εδώ πιστεύω ότι υπάρχει πεδίο βελτίωσης των σχέσεων, διότι οι αποστολές αυτές έχουν πόρους αποτελεσματικούς και αυτή τη στιγμή έχουν και συγκεκριμένα αποτελέσματα επί των εκλογών. Όμω υπάρχουν και συγκεκριμένες προϋποθέσεις και συστάσει που πρέπει να τηρούνται και συμφωνώ με, ότι με τους πόρους που έχει το μέσον αυτή τη στιγμή δεν είχαμε τη δυνατότητα να προωθήσουμε αυτές τις σχέσει. και γι' αυτό πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο για να αντιμετωπίσουμε και το θέμα το οποίο συστήξατε. Προς την κυρία Γέγκλε, σχετικά με την ανάπτυξη της υπαίθρου. Ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Πιστεύω ότι αυτό εξηγεί πολύ καλά τη συμπληρωματικότητα αυτού του μέσου. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Στην Τανζανία Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη, για να μπορέσει η χώρα να βελτιώσει την ε, αγροτική παραγωγή της. Εδώ θα μπορούσε να υπάρξει κάποια επίπτωση στα ανθρώπινα δικαιώματα σχετικά με τα δικαιώματα που έχουν ε, επί αγροτικών περιοχών κλπ. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι διαχωρίζουμε ε, τα μέσα, αλλά θα ήταν ε, εσφαλμένη αυτή η αντιμετώπιση, το να διαχωρίσουμε δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα από την αγροτική ανάπτυξη. Και γι' αυτό λέμε ότι τέτοιου είδους θέματα θα πρέπει ε, να αντιμετωπίζονται με ενιαίο τρόπο. Δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα να μπαίνουν ε, μέσα στα θέματα ανάπτυξης, να μην χρησιμοποιούμε το μέσο χωριστά. Και σε άλλες χώρες έχουμε ε, αντίστοιχες περιπτώσεις. Προς την κυρία Βάιντερε που ρώτησε για το μηχανισμό και για την άμεση χρηματοδότηση. Όντως, είναι δύσκολο θέμα οι αιτήσει χρηματοδότηση. Όχι μόνο για το μέσο ΕΜΔΑ όμω, για όλα τα μέσα οι αιτήσει χρηματοδότηση είναι μια δύσκολη διαδικασία και εδώ είναι περισσότερο ευάλωτοι αυτοί οι οποίοι θα κάνουν αιτήσει χρηματοδότηση. Θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τη διαδικασία και θα προσπαθήσουμε να, διατηρούμε, να τηρούμε όλου ενήμερου. Προ τον κύριο Χάουιτ που σίγουρα το πνεύμα του μας συνοδεύει στην απάντηση που του δίνω τώρα. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη που μας δίνετε για την αποδέσμευση του μέσου και για τους υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα βρούμε τον τρόπο να σας ενημερώνουμε εμπιστευτικά για τα όσα κάνουμε. Για τους ομοφιλόφιλους ε, και διαφιλικούς ε, Υπάρχει σε ένα σημείο στο κείμενο, στο 3β, δεύτερο εδάφιο, αν δεν είναι αρκετά ε, επαρκής η διατύπωση μπορούμε να το βελτιώσουμε. Και νομίζω ότι είναι θέμα διατύπωσης. Για τις κατεξουσιοδότηση πράξης τώρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα και η Πρόεδρος της Επιτροπής νομίζω τόνισε πόσο σημαντικό είναι. Ο λόγος για τον οποίο δεν το βλέπετε σε αυτόν τον κανονισμό είναι ότι το χειριζόμαστε στον οριζόντιο κανονισμό. Μην νομίζετε λοιπόν ότι, έχουν, ότι αγνοεί η, Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη συμφωνία που έχει γίνει. Απλώς προτείνουμε να το αντιμετωπίσουμε συνολικά μέσω του κοινού κανονισμού εφαρμογής. Μια απάντηση προς την κυρία Γκόμες. Καταρχήν, η ίδια απάντηση όσον αφορά τι κατεξουσιοδότηση πράξη, και εσείς ρωτήσατε συγκεκριμένα για την Αιθιοπία και τι σχέσει με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη. Επανέρχομαι στην απάντηση που έδωσα για τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Εδώ πρέπει να δείτε το μέσο ΕΜΔΑ ολιστικά, σφαιρικά, μέσα στο πλαίσιο δηλαδή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη χώρα αυτή συνολικά. για το αν υποστηρίζουμε τις πληρωμές, για το αν η Αιθιοπία αξίζει να υποστηρίξουμε τον προϋπολογισμό ότι αν πρέπει να δουλεύουμε με μη κυβερνητικέ οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς. Έτσι ξεκίνησα την παρουσίασή μου. Είπα ότι είναι κατάλληλη η χρονική στιγμή για να υποστηρίξουμε περισσότερα τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η διεθνής κατάσταση παρότι το Ταμείο για την Ανάπτυξη δεν εκφράζεται ως προϋπολογισμός, νομίζω ότι ακριβώς αυτή η σφαιρική προσέγγιση μας βοηθάει να συνδυάσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις ε, ανησυχίες μας για την ανάπτυξη. Ρωτήσατε και για τη Λιβύη. Ήδη υποστηρίζουμε σήμερα την εκπόνηση του εκλογικού νόμου στη Λιβύη και το επόμενο βήμα θα είναι η εκπαίδευση που θα παρέχουμε προς τα πολιτικά κόμματα. δεν δίνουμε άμεση υποστήριξη σε ένα πολιτικό κόμμα για μικροκομματικούς σκοπούς. Απλώς υποστηρίζουμε τη Λιβύη με την σύνταξη του εκλογικού νόμου και με κατάρτιση που παρέχουμε στα εκλογικά κόμματα και θα υποστηρίξουμε και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στη Λιβύη που θα φροντίζουν για την υλοποίηση αυτών των δημοκρατικών κανόνων. Προς τον κύριο Μακμίλαν Σκότ θέλω να πω ότι συμφωνώ μαζί σας. Υπάρχει υψηλή υποστήριξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ισχυρή πολιτική υποστήριξη και γι' αυτό προτείνει η Επιτροπή 4% αύξηση αυτού του μέσου. Και πρέπει να σας πω ότι όταν υπογράφω αυτά τα έγγραφα επιχορηγήσεων των 10.000 ευρώ, είναι αυτή η μία στιγμή, μία μέρα την εβδομάδα που υπογράφω αυτά τα έγγραφα, που είναι πολύ δύσκολη, γιατί ξέρω ότι κάποιους ε, βοηθάμε, αλλά δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε όλους. Ήδη έχουμε ε, στο χαρτοφυλάκιο των άμεσων αυτών ε, επιχορηγήσεων γύρω στα 50 έργα και έχουμε άλλα 50 τα οποία επίκυνται. Και θα σας ενημερώνουμε ατύπως για τις δράσεις μας με αυτά τα ε, κονδύλια, με αυτές τις άμεσες επιχορηγήσεις. Περνάω τώρα σε ένα σχόλιο που κάνατε ότι το παρελθόν το μέσον ήταν περισσότερο εργαλείο ανάπτυξης και όχι τόσο εργαλείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι συζητήσιμο αυτό το θέμα. Εμείς θα θέλαμε να είναι ένα εργαλείο για τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα εστιάζει σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σαφώς. Ίσως έχετε δίκιο ότι κάπως ξεφύγαμε με την υποστήριξη οργανώσεων κοινωνίας των πολιτών που δεν αποσκοπούσαν καθαρά σε δράσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα έλεγα ότι μεγαλύτερο πρόβλημα θα ήταν ε, ε, να μας προτείνεται να χρησιμοποιήσουμε τα κονδύλια για να υποστηρίξουμε διεθνείς οργανισμούς. Παρότι πολλοί από αυτούς ε, είναι κλειδιά για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γιατί αν τα περισσότερα κονδύλια μας τα, τα δώσουμε για να χρηματοδοτήσουμε οργανώσεις του ΟΗΕ θα είναι μεν σημαντικό, αλλά εμείς έχουμε να κάνουμε και κάτι παραπάνω για να υποστηρίξουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και προς την Πρόεδρο, σχετικά με τους ενδογενείς πληθυσμούς, όχι δεν είναι τέτοια η πρόθεσή μας, δεν έχουμε την πρόθεση να μειώσουμε τις δράσεις μας σε αυτό το τομέα. Αυτά διότι έχω μακρηγορήσει. Ο Πατρίς συνεχίζει να μου δίνει σημειώματα, αλλά άμα έχω ξεχάσει κάτι, θα ζητήσω από τον Πατρίς να τα πει ο ίδιος. Πολύ σύντομα, εγώ θέλω να απαντήσω για την ευελιξία. Τέσσερα σημεία. Πρώτον, η ανάγκη μεγαλύτερη απλούστευσης ε, του κανονισμού είναι κάτι που τόνισε και ο πρόεδρος Μπαρόζο. Αυτό ισχύει λοιπόν για όλα τα μέσα ε, Εμεί έχουμε δουλέψει τα τελευταία δύο χρόνια με την κοινωνία των πολιτών και με το διαφρομένο διάλογο, προσπαθώντας να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω. Αποκινούμε την κοινωνία των πολιτών για να αντιμετωπίσουμε διάφορα ζητήματα. Και ένα από αυτά τα ζητήματα είναι μια απλουστευμένη διαδικασία στα καθημερινά ζητήματα. Δουλεύουμε λοιπόν πάνω σε τέτοια ζητήματα. Ε, δεύτερον, το θέμα τη εκπαίδευση και κατάρτιση είναι πολύ σημαντικό και κάθε χρόνο κάνουμε μια συνάντηση ετήσια με τι μη κυβερνητικέ οργανώσει για να αποφασίσουμε πώ μπορούμε να τι βοηθήσουμε καλύτερα. Το ίδιο κάνουμε και με τι δικέ μα αντιπροσωπείε για να μπορούν οι αντιπροσωπείε μα να αντιμετωπίζουν προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία των πολιτών επιτόπου. Τρίτον, προσπαθούμε να εξετάζουμε όχι τα βήματα τη διαδικασία, αλλά τα έντυπα που χρησιμοποιούνται, τους μορφότυπους που χρησιμοποιούνται για να απλουστεύσουμε τη διαδικασία ε, ε, υποβολής αιτήσεων. Όταν ε, θα έχουμε ολοκληρώσει το δημοσιονομικό κανονισμό θα είναι μεγαλύτερη απλούστευση προς όφελος όλων. όταν εγκριθεί ο χρηματοδοτικός κανονισμός. Και τέλος, για, την, για το μέσο που προτείνουμε, για τη διευκόλυνση, είναι κάτι το οποίο θα χρησιμοποιούμε, όπως είπε ο Κριστιαν, για την Συρία. Είναι κάτι που θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα και να έχουμε αποτελέσματα γρήγορα. Είναι ένα μέσο διευκόλυνσης που μας παρέχεται. Καταλαβαίνουμε την απογοήτευση της κοινωνίας των πολιτών ε, σε πολλές περιπτώσεις, αλλά είναι πολύ ανταγωνιστική η κατάσταση. Ο προπολογισμό είναι μικρός ε, και μόνο με περισσότερα χρήματα θα μπορούσαμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους δυο σας για τις απαντήσεις σας. Πριν ε, δώσω τον λόγο στον κύριο Τίμαν, να σας υπενθυμίσω ως... έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Θα ήθελα να ξεκινήσω την ώρα των ερωτήσεων στις 11 και μετά υπάρχει και ο εισηγητής να μιλήσει. Κύριε Τίμαντς, κυρία Πρόεδρε, συγχαρητήρια και από μένα για την επανεκλογή σας και στους αντιπρόεδρους επίσης και στον κύριο Λάμπστορφ ε, επίσης ε, για το ότι είναι εισηγητής. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος γιατί νομίζω πως ο κύριος Σμιτ ήταν αρκετά αναλυτικός. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα και επειδή πρόκειται πρώτα απ' όλα για ένα θεματικό μέσο να πω τα υπενθυμίσω τα εξής είναι σημαντικό να αντιληφθούμε πως ε, το νέο αυτό μέσο, το ΕΜΔΑ, έχει μόνο 8 άρθρα, ενώ πριν είχε 21, οπότε περιορίζεται, είναι ένα θεματικό μέσο. Αλλά σημαντικό είναι να δούμε το σχέδιο κανονισμού για τις κοινέ διαδικασίες πως προβλέπει δύο σημαντικά άρθρα όσον αφορά την εφαρμογή σε σχέση με το ΕΜΔΑ, το άρθρο 6 και το άρθρο 11. Το άρθρο 11 αφορά τον ε, κύκλο των ε, δικαιούχων, την επιλεξιμότητα και το άρθρο 11 προβλέπει την ε, διαδικασία Ε, εκταμίευσης. Ε, το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να πω είναι πως προσπαθήσαμε στη διαμόρφωση αυτού του μέσου να επιφέρουμε κάποιες συμπληρώσεις ιδιαίτερα στην παράγραφο 2, δηλαδή στο άρθρο 2 όσον αφορά δηλαδή το πεδίο εφαρμογής ε, ε, υπάρχει μια ειδική ρήτρα για την ε, ελευθερία την θρησκευτική που αφορά εξελίξεις παραδείγματος χάρη στην Ιγυρία, το Πακιστάν ε, και αλλού που είναι για εμάς ιδιαίτερα σημαντικό. Υπάρχει επίσης και η παράγραφος για την ελευθερία γνώμης και ΜΜΕ που αναδιατυπώθηκε και εκεί πέρα αναφέραμε ειδικά την ελευθερία του διαδικτύου. Και αυτό αφορά το ερώτημα του κυρίου Χάουιτ. Ρητά δε τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα και τα πολιτιστικά καθώς επίσης και την εταιρική κοινωνική ευθύνη που μας απασχολεί ιδιαίτερα. Αυτό το οποίο θα ήθελα επιπλέον να πω είναι πως είναι πως θεωρούμε πως ο δομημένος διάλογος των προηγούμενων ετών μεταξύ Κομισιόν και Κοινοβουλίου πρέπει να συνεχιστεί, το υποστηρίζουμε πλήρως θεωρούμε πως η συμπερίληψη του Κοινοβουλίου είναι σημαντική. Επίσης θεωρούμε πως είναι σημαντικό να απλοποιηθεί η εφαρμογή των έργων, ειδικά όταν μιλάμε για τοπική δημοσίευση των, ε, της ε, πρόσκλησης υποβολής ε, προσφορών, τυχόν διαγωνισμών δηλαδή, θα πρέπει να φροντίσουμε οι τοπικές μήκυο να έχουν καλύτερη πρόσβαση. Και το τελευταίο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι το εξής. Και στο μέλλον, υπό το μέσο αυτό, θα χρηματοδοτούνται οι παρατηρητές των εκλογών από αυτό το μέσο και πρέπει να διασφαλίσουμε πως ο συμβιβασμός ο οποίος βρέθηκε το 2006, ότι δηλαδή θα υπάρχει ένα maximum 25% για παρατήρηση εκλογών, δεν θα πρέπει να ξεπεραστεί για να υπάρχει ισορροπία μεταξύ χρηματοδότησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων αφενός και παρατήρησης ε, εκλογών αφετέρου και να μην διαταραχθεί. Αυτά ήταν τα ε, ζητήματα αυτά που μας απασχολούν ιδιαίτερα στην ε, υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ε, αλλιώς επιβεβαιώνω πως συνεργαζόμαστε στενά με τους συναδέλφους της Κομισιόν και οπωσδήποτε θα προσπαθήσουμε και στις διαπραγματεύσεις που έχουμε και με το Συμβούλιο και με το Κοινοβούλιο να έχουμε μια κοινή κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Λάμζορφ. Ναι, δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Ήταν αρκετά μακροσκελής η συζήτηση και νομίζω είναι σαφές και από αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι το που δίνουμε εμείς βάρος. Χαίρομαι για το ότι έχουμε τώρα και την ελευθερία του ίντερνετ αλλά δεν άκουσα στις απαντήσεις της Κομισιόν και τις υπηρεσίες εξωτερικής δράσης. Μια απάντηση για το ερώτημα του κυρίου Χάουιτ για τα ζητήματα ΛΟΑΤ. Κάτι άλλο που είπε η Άννα για τις πράξεις κατ' εξουσιοδότηση. Στην πολιτική γειτονία αυτό αναφέρεται ρητός, δηλαδή υπάρχει ε, όχι οριζόντια, αλλά αναφέρεται στο ίδιο το κείμενο. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι είναι λογικό και πώς θέλουμε να το γράψουμε. Ένα από τα πιο δύσκολα και πιο ακαθόδη ζητήματα, αλλά και οπωσδήποτε πιο ενδιαφέροντα, θα είναι το θέμα της δημοκρατίας, το δέλτα στο ΕΜΔΑ και το πώς θα μπορέσει να υπάρξει ένας διαχωρισμός. Μιλήσατε αφενός για πλουραλισμό κτλ. Από την άλλη, το e ίδιο αυτό το οποίο προωθεί και η Πολωνική Προεδρία ε, είναι κάτι διαφορετικό βεβαίως. Θα να βρεθεί το όριο θα είναι κάπως δύσκολο, όπως είπε και ο κύριος Χάβιτ έχει κάποιο δίκαιο, δηλαδή τι είναι κόμμα και τι δεν είναι κόμμα. Αλλά είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει και προς όφελος των ε, δικαιούχων αλλά και των φορολογούμενών μας. Επίσης να διορθώσω την παράληψή μου, την ασυγχώρητη, να σας συγχαρώ και εγώ κυρία Πρόεδρε. Ε, πράγματι, κύριε Λάμσδορφ, είναι καλό το ότι έχουμε ε, εισηγητή για αυτό το θέμα κάποιον ο οποίος το παίρνει ε, σοβαρά. Και είναι σημαντικό το ότι είστε από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και οι προηγούμενοι εισηγητές ήταν από αυτή την Επιτροπή και είναι καλό το ότι υπάρχει τώρα αυτός ο δομημένος διάλογος όπως είπε ο Ρίτσαρτ. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ομάδα για την ΕΜΤΑ η οποία θα συνεχίσει το έργο της. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω τις διάφορες πολιτικές ομάδες να μου πούν ε, ποιοι βουλευτές ασχολούνται με αυτό και έτσι ώστε να συναντηθούμε στην επόμενη ολομέλεια του Στρασβούργου. να συζητήσουμε το ετήσιο πρόγραμμα δράσης, αλλά και σε εσάς κύριε Σμίτ που είπατε πως πρέπει να βρεθεί ε, ένας τρόπος για να μην ε, λέμε δημόσια το ποια έργα θα στηρίξουμε. Ε, πάντα αυτή την ομάδα εργασίας χρησιμοποιούμε που συνεδριάζει και κλεισμένων των θυρών. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους για την ουσιαστική αυτή συζήτηση και πρέπει να πω πως ε, ξεπεράσαμε τώρα το χρόνο μας και τώρα προτείνω να γίνει το εξής στην ώρα των ερωτήσεων. Υπάρχουν οι ερωτήσεις στα έγγραφά σας, ο κάθε βουλευτής ξέρει τι ρώτησε, οπότε θα αναφέρω μόνο τον τίτλο και θα παρακαλέσω την Κομισιόν να απαντήσει. Πρώτη ερώτηση είναι του κυρίου Ταβάρες και αναφέρεται σε έναν νόμο στο Ισραήλ για την παράνομη μετανάστευση. Παρακαλώ να απαντήσετε. Ποιος θα δώσει την απάντηση. Ορίστε. Ο κύριος Σουάν. Παρακαλώ. Α, διάστηκα, με συγχωρείτε.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 Με συγχωρείτε που ήρθα τελευταία στιγμή. Υπήρχε ένας συνάδελφος που θα απαντούσε σε αυτή την ερώτηση. Με την άδεια του κυρίου Ταβάρες έχετε μια, αν έχετε μια άλλη ερώτηση να απαντήσετε, να απαντήσετε σε αυτήν και θα περιμένουμε τον συνάδελφό σας. Είχαμε πει ότι θα αρχίσουμε και 11 παρά. Κύριε Σουάν, ποια ερώτηση μπορείτε να απαντήσετε. Μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση για την Ουκρανία. Μάλιστα. Ε, καλημέρα σας. Είμαι ο υπεύθυνο για την Ουκρανία στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ε, παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην Ουκρανία. Είπα ότι η εκπρόσωπος της είπα της εκπροσώπου εξέφρασε την ισχύα της για το ότι δεν αντιμετωπίστηκαν σωστά οι ελλείψεις στην ε, πρώτη δίκη της Ιουλίας Τιμοσένκο για την οποία ξέρετε πως θέση μας ήταν πως δεν είχε διεξαχθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά την δίκαιη δίκη. Η κυρία Τιμοσένκο που είναι η σημαντική μορφή της αντιπολίτευσης δεν μπορεί τώρα να κατέβει σε επόμενε βουλευτικέ εκλογέ. Πολλέ άλλε ε, Πολλοί άλλοι αντιπολιτευσής επίσης δεν θα μπορέσουν να το κάνουν και είναι ε, λυπηρό το ότι πρέπει να ασχολούμαστε με ζητήματα δικαιοσύνης στην Ουκρανία. Όσον αφορά τώρα το ερώτημα το πώ επηρεάζουν οι εξελίξει στην Ουκρανία τι διαπραγματεύσει ε, για τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Κοιτάξτε, συνεχίστηκαν τεχνικές διαπραγματεύσεις για την συμφωνία αυτή, για τη σύσταση μιας ε, περιοχής ε, ελευθέρου εμπορίου με την Ουκρανία. Με στόχο να ολοκληρωθεί η συμφωνία όπως ε, ζήτησαν και πάρα πολλές ε, ΜΚΟ και οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών. Ταυτόχρονα η κοινή δήλωση της Συνόδου Κορυφής 19 Δεκεμβρίου με την ε, Ουκρανία ανέφερε σαφώς πως ο σεβασμός του κράτους και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ταχύτητα της ε, ενσωμάτωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και της ισχύω της συμφωνίας και της εφαρμογής της. Επίσης, στην ερώτηση αναφέρατε οι αστυνομικές ε, αυθαιρεσίες στην Ουκρανία. Η άποψή μας είναι πως πράγματι πρέπει να ενισχυθεί η νομοθεσία περί ελευθερίας του συνέρχεστα στην Ουκρανία γιατί όταν γίνεται μία διαδήλωση στην ε, Ουκρανία δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες για την παρέμβαση της αστυνομίας και αυτό οδηγεί σε συχνές περιπτώσεις υπερβολικής ε, βίας ε, κατά ειρηνικών διαδηλωτών. Επιπλέον αναμένουμε από τις αρχές να εξετάσουν προσεκτικά τυχόν αναφορές για αστυνομικές αυθαιρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα. Ε, σας διαβεβαιώ πως ε, θίγουμε αυτά τα ζητήματα στις διμερείς επαφές μας με την Ουκρανία και ευχαρίστω ε, να σας ενημερώσουμε όποτε θέλετε για τις εξελίξεις. Μάλιστα, δεν νομίζω να υπάρχει συμπληρωματική ερώτηση. Βλέπω πως η Φρίντα Μπρέπουλς απουσιάζει. Μπορούμε λοιπόν να πάμε στο ερώτημα της Νικόλ Κιλ Νίλσεν για την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερβαϊτζάν. Μπορείτε να μας απαντήσετε γι' αυτό. Κοιτάξτε, θα κάνουμε το εξής, κύριε Σβάν. Έχουμε πέντε ερωτήσεις. Ε, ποιες μπορείτε να μας απαντήσετε. Ε, με, με συγχωρείτε. Είχα κανονίσει να έρθουν άλλοι συνάδελφοι να απαντήσουν στις ερωτήσεις θα επιληφθώ του θέματος μετά από τη συνεδρίαση οπωσδήποτε. Ε, έχω κάποιο συνάλφο που μπορεί να απαντήσει για την Αιθιοπία, εν πάση περιπτώσει. Είναι και ένα γκόμες εδώ. Να ακούσουμε λοιπόν. Λοιπόν, το θέμα, η ερώτηση αφορά την Αιθιοπία και θα ήθελα να μας απαντήσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τόμας Χάντελ, από το Γραφείο για την Αιθιοπία στο Τμήμα Αφρικής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερική Δράσης. Το ερώτημα έχει σχέση με την κατάσταση στην Αιθιοπία και συγκεκριμένα ε, σχετικά με δύο Σουηδούς δημοσιογράφους που καταδικάστηκαν σε 11 χρόνια φυλάκισης ε, ε, κατηγορούμενοι για τρομοκρατία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η Επιτροπή παρακολουθούν το θέμα αυτό και το Δεκέμβριο, την ημερομηνία της καταδίκης τους, η κυρία Άστον έκανε μια δήλωση όπου εκφράζει ανησυχία για την εφαρμογή του αντιτρομοκρατικού νόμου και εκφράζει την ελπίδα ότι οι δύο Σουηδοί δημοσιογράφοι, καθώς και δημοσιογράφοι από την Αιθιοπία που κατηγορούνται βάσει του ίδιου νόμου, θα απελευθερωθούν. Όσον αφορά το Μάρτιν Τσκίπρο και το Γιώχαν Πρέσον, υπάρχει τώρα μια νέα εξέλιξη, γιατί έχουν αποδεχθεί την καταδίκη τους και αφού απεδέχθησαν την ετοιμιγορία, κλείνει η νομική διαδικασία στην Αιθιοπία. Το παρακολουθούμε το θέμα σε συντονισμό με την κυβέρνηση της Σουηδίας. Και στο παρασκήνιο γίνονται τώρα οι εξελίξεις. Εμείς τώρα παρακολουθούμε το τι γίνεται με την κυβέρνηση της Σουηδίας που θεωρεί ότι με τη διπλωματία θα επιλύσει αυτό το θέμα και προσπαθούν να επιτύχουν την απελευθέρωσή τους δια της διπλωματικής οδού. Η υπόθεση των δύο Σουηδών δημοσιογράφων ήταν η πρώτη υπόθεση στην οποία είχαμε μία δίκη βάσει του αντιτρομοκρατικού νόμου που θέσπισε η Αιθιοπία το 2009. Θεωρήθηκαν ένοχοι αλλά η ερμηνεία για την τρομοκρατία είναι αυτό που μας ενδιαφέρει στη συγκεκριμένη περίπτωση για το τι σημαίνει τρομοκρατία. Σίγουρα σχετίζεται με τον περιορισμό της ελεύθερης έκφρασης και, και των μέσων ενημέρωσης. Υπάρχει απειλή τρομοκρατίας στην Αιθιοπία και η πρόσφατη επίθεση σε τουρίστες στη Βόρεια Ιθιοπία είναι ένα παράδειγμα αυτών των τρομοκρατικών δράσεων. Επομένως, η Αιθιοπία καταλαβαίνουμε ότι θέλει να καταπολεμήσει την τρομοκρατία. Όμως αυτή η καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν πρέπει να αποτελέσει μέσο για την ε, καταπίεση των πολιτικών αντιφρονούντων. Ζητήσαμε λοιπόν επισήμω από την κυβέρνηση με βάση το άρθρο 8 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον πολιτικό διάλογο για την ελευθερία του τύπου και την εφαρμογή του αντιτρομοκρατικού νόμου. Το δεύτερο μέρος της ερώτησής σας αφορούσε την ε, αναπτυξιακή βοήθεια στην Αιθιοπία και ε, ε, την Συμφωνία Κοτονού και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συνεχίζουμε το διάλογο μας με την Αιθιοπία. Υπάρχει μια μακρά εταιρική σχέση με την Αιθιοπία. Και όπως σας είπα, το παρακολουθούμε αυτό το θέμα και βάσει του πολιτικού διαλόγου, βάσει του άρθρου 8, Είμαστε σε συνεχείς συζητήσει. Το έχουμε ζητήσει από την Αθιοπία. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκόμες, χωρίς μικρόφωνο. Μία μακρά εταιρική σχέση με ένα καθεστώς ε, ε, που καταπιέζει ένα καθεστώς που καταπιέζει το λαό του. που τώρα, και όχι μάλλον τώρα, πολύ καιρό τώρα, αλλά τώρα υπάρχει και σε νόμο, τώρα κατέφυγε στην χρήση της έννοιας της τρομοκρατίας με καταχρηστικό τρόπο για να μπορέσει ε, να καταπιέσει και αιθίωπες πολίτες και αλλοδαπούς που τολμούν να μιλήσουν κατά της ε, βίας. Αυτή η διακριτική προσέγγιση που ακολουθείτε δεν νομίζω ότι θα έχει αποτέλεσμα. Μακάρι να έχει αποτέλεσμα, αλλά φοβούμαι ότι δεν θα έχει. Και θα ήθελα να ρωτήσω αυτοί οι δύο δημοσιογράφοι γιατί δέχτηκαν την ετοιμιγορία, γιατί δέχτηκαν ότι είναι ένοχοι. παρακολουθούσε τη δίκη κάποιος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, του συμβούλευσε κάποιος να το κάνουν. Γιατί ξέρω ότι υπάρχει μια τέτοια παράδοση στην Αιθιοπία. Όντω δηλώνουν ότι είναι ένοχοι για οτιδήποτε. Αυτό είχε γίνει και τον ε, Ουμπέρτο Κανεντάξη, ένα πρώην μέλο κόμματο τη αντιπολίτευση που είχε φυλακιστεί ισοβίω και δήλωσε δύο φορές ένοχη, αποδέχεται την ενοχή της για να μπορέσει να λάβει χάρη και να απελευθερωθεί. Υπάρχει όμως κάποιος σύμβουλος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την αντιπροσωπεία, είτε κάποιος γνωστός ε, σύμβουλος στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που του συμβούλευσε να δεχθούν αυτή την ετοιμιγορία. Ευχαριστώ κυρία Γκομές. Μπορείτε να μας απαντήσετε. Ευχαριστώ. Η, Ευρω... η αντιπροσωπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και οι Ηνωμένε Πολιτείες ε, παρακολουθούσαν τη δίκη. Είχαν Σουηδούς δικηγόρους, οι δύο Σουηδοί δημοσιογράφοι. Υπήρχαν και μάρτυρες από ολόκληρο τον κόσμο που μίλησαν, που έλεγαν το λόγο υπέρ τους, κατέθεσαν υπέρ των δύο Σουηδών δημοσιογράφων. Δεν ξέρω ποιοι ήταν οι λόγοι που τους οδήγησαν να μην ασκήσουν έφεση αλλά να δεχθούν την ετοιμιγορία. Ευχαριστούμε πολύ. Και έχω μια πρόταση για τις άλλες ερωτήσεις ή μήπως, μήπως έχει έρθει κανείς που μπορεί να απαντήσει, κύριε Σουάν. Ξέρετε, η Επιτροπή είναι ένα ένας με χιλιάδες ε, πρόσωπα και έρχεται ο συνάδελφος από ό,τι μου λένε να απαντήσει για το Ισραήλ. Εγώ μπορώ συνοπτικά να απαντήσω για τις Ηνωμένε Πολιτείε και για το νόμο των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την εθνική άμυνα. Αν σας εξυπηρετεί η δική μου απάντηση. So I think, um, um... The colleague of Frida Πρόεδρος, νομίζω ότι η συνάδελφος της Φρίντα Beavers και ε, η Νικόλ Κιλ θα παρακολουθήσουν την απάντηση στην ερώτηση της Φρίντα. Κύριε Σουάν, έχετε τον λόγο. Okay, sorry, I was um, expecting the, the, the question first, but... Uh... Λοιπόν, για το θέμα αυτού του νόμου για την εθνική άμυνα στι ΗΠΑ, θέλω να πω ότι αυτή η νομοθεσία είναι συμβατή με τι διεθνεί υποχρεώσει και οι επιπτώσει επί των συμφωνιών Ευρωπαϊκή Ένωση ΗΠΑ αναλύεται προσεκτικά, ιδιαίτερα στα θέματα που δεν καλύπτονται από τη δήλωση του Προέδρου Ομπάμα, μεταξύ άλλων, και για το αν οι πήκοοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ύποπτοι για τρομοκρατία μπορούν να θεωρηθούν ύποπτοι και να καταδικαστούν χωρί δίκη να κρατούνται χωρί δίκη και συζητούνται τα θέματα αυτά με τις Αμερικανικές αρχές. Αν δεν υπάρχει κάποια συνέχεια στην ερώτηση, ας προχωρήσουμε γιατί έχουμε υπερβεί το χρόνο μας. Α, βλέπω ότι η κυρία Κιλ Νίλσεν έχει κάποια ερώτηση. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη γιατί πρέπει να αποχωρήσω, αλλά έχω μια ερώτηση για το Αζερβαϊτζάν αν έρθει κανείς για να απαντήσει στην ερώτησή μου, θέλω να προσθέσω ένα σημείο που το θεωρώ σημαντικό γιατί είναι πάρα πολύ επίκαιρο. Ο ειδικό εισηγητής για τους πολιτικούς κρατουμένους στο Αζερμπαϊτζάν, ο ειδικό εκπρόσωπος από το Συμβούλιο, από τη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου τη Ευρώπη, για το, το είναι μέλο του Συμβουλίου τη Ευρώπη, ο ειδικό εισηγητή δεν μπορεί, και αυτό είναι εντελώ νέο, είναι σημερινό θέμα, δεν μπορεί να πάρει βίζα θεώρηση διαβατηρίου για να πάει στο Αζερβαϊτζάν. Το προσθέτω λοιπόν αυτό στην ερώτησή μου που ήδη έχω κάνει σχετικά με τον περιορισμό της ελευθερίας έκφρασης στο Αζερβαϊτζάν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα μπορούσε ο συνάδελφος να απαντήσει στις ερωτήσεις όταν θα περάσουμε στα διάφορα. Αν δεν είναι δυνατό να γίνει αυτό, θα είναι το πρώτο σημείο στην απογευματινή συνεδρίαση. Διαφορετικά, θα συζητήσουμε μια γραπτή απάντηση στην ερώτηση. Θα σα ζητήσουμε να στείλετε την απάντηση στο βουλευτή που, άσκησε, που έκανε την ερώτηση με αντίγραφο στη γραμματεία της Υποεπιτροπής Ντρουά γιατί μας ενδιαφέρουν όλους οι απαντήσεις σας. Και ελπίζω ότι την επόμενη φορά δεν θα υπάρξει τέτοια παρανόηση και θα υπάρχουν αυτοί που πρέπει να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Γιατί πάντοτε υπάρχει δυσκολία στο ε, να βρίσκονται εδώ οι ευρωβουλευτέ που έχουν κάνει τι ερωτήσει στην κατάλληλη χρονική στιγμή. Και τώρα θα ήθελα να καλωσορίσω ένα νέο μέλο στην Επιτροπή Ντροά, τον κύριο Μπροκ. Κύριε Μπροκ, έχετε ένα πράσινο ταμπελάκι ως αναπληρωτής ε, στην Επιτροπή Τρουάς. Σας καλωσορίζω λοιπόν ε, ως μέλος της ΑΦΕΤ. Θα ξεκινήσουμε στις 11.30 με το διευρυμένο Προεδρείο. Αν θέλετε, μείνετε. Με μεγάλη μας χαρά θα σας έχουμε κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Απλώς ε, ήρθα για να δείξω ότι πραγματικά έχω ενδιαφέρον για τις εργασίες αυτής της υποεπιτροπής και με μεγάλη χαρά ε, θα συνεργαστώ ε, και με το Διευρυμένο Προεδρείο και τις επόμενες εβδομάδες σε συνεργασία με το σύνολο της Επιτροπής. για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας ε, για τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για το ρόλο το, της ρήτας ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εμπορικέ πολιτικές για να μπορέσει να γίνει περισσότερο λειτουργικός ο ρόλος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι θέματα στα οποία η δική σας υποεπιτροπή έχει ε, τον κύριο ρόλο. Αυτό ήθελα απλώς να τονίσω. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. Είχαμε πολλούς βουλευτές παρόντες σήμερα γιατί συζητήσαμε το θέμα του μέσου ΕΜΔΑ. Χαίρομαι ιδιαίτερως ε, που αφιερώνετε χρόνο στο να έρθετε εδώ εσείς ως πρόεδρος της ΑΦΕΤ σε αυτή την υποεπιτροπή. Ε, δεν υπάρχουν διαφορές απόψεων με την ΑΦΕΤ, αλλά είναι καλό να έχουμε την υποστήριξή σας για τα ψηφίσματα τα οποία προετοιμάζουμε εδώ, τα οποία πολλές φορές θέλουμε να περνούν από την ΑΦΕΤ. Και χαιρόμαστε για μια αύξηση των δυνατοτήτων, ώστε να έχουμε διευρυμένο διευρυμένη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να μπορούμε να έχουμε συμφωνία στα διάφορα θέματα με ευρεία συνένεση. Και όταν έχουμε ε, γνωμοδοτήσει πρωτοβουλίε και όταν έχουμε προσκεκλημένους εμπειρογνώμονε και όταν κάνουμε μελέτες, καλό είναι να αλληλοσυμπληρωνόμαστε και να γίνονται όλα αυτά με συντονισμένο τρόπο. Και άλλη μια φορά σας ευχαριστώ. Και αν θέλετε, περιμένετε λίγο, θα αρχίσει στις 11.30 το διευρυμένο Προεδρείο και προς όλους τους άλλους συναδέλφους και τα υπόλοιπα μέλη του προσωπικού, θα ήθελα να πω ότι θα είναι και κλεισμένων των θυρών η συνεδρίαση του Διευρυμένου Προεδρίου. Θα ξεκινήσουμε το απόγευμα με την ακρόαση για το Διαμερικανικό Μηχανισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.